Dear colleagues, good morning. Καλημέρα συνάδελφοι, είναι ώρα να ξεκινήσουμε την συνεδρίασή μας. Βρισκόμαστε πλέον στο σημείο, παρακαλώ. Sorry about this chair, but I... Συγγνώμη Πρόεδρε, αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Ε, μια και η υπερβάωση είναι εδώ, να πω ότι λάβαμε την εκδοχή της, ε, ε, στις, ε, στις 2.30 τον κατάλογο ψηφοφορίας για την έκθεση Μπερές που είναι 57, συγγνώμη, 75 σελίδες. Δεν είναι σωστός τρόπος εργασίας αυτός. Δεν είχα καν την ευκαιρία να ελέγξω και επομένως δεν νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε σήμερα γιατί ε, όταν σε μια τόσο σημαντική έκθεση λαμβάνουμε την, ε, ε, τον κατάλογο ψηφοφορία στην τελευταία στιγμή που είναι και τόσο μεγάλος δεν είναι συνθήκες αυτές και δεν μπορώ να αναλάβω την, ε, την ευθύνη της ψηφοφορίας. Δεν θα έχω το χρόνο να συζητήσω με τους συναδέλφους. Ζητώ λοιπόν να μην εγγραφεί το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη στην ώρα της ψηφοφορίας. Πρόεδρος, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά Εξ όσων γνωρίζω, είχαν κυκλοφορήσει ήδη εδώ και πολύ καιρό οι συμβαστικές ε, λύσεις ε, στο τελευταίο κατάλογο ψηφοφορίας ε, είναι ε, πολύ λίγα τα καινούργια πράγματα. Στην ουσία η σειρά των τροπολογιών και το τι καλύπτεται κάθε φορά. Γι' αυτό νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε ακόμα απαρτία και επομένως θα πρέπει να συνεχίσουμε. Και μετά, μετά μπορείτε να ξαναθίξετε το ζήτημα αυτό, να το εγείρετε εν ευθέτω χρόνο. Είναι δικιά σας απόφαση κύριε Πρόεδρε ε, λέει ο κύριος Γκίγκολτ. Και βεβαίως εσείς λέτε ότι απλώς εδώ η διαφορά είναι τι καλύπτεται και τι όχι, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία καλύπτονται ή όχι και τα οποία ε, θα, πληρω... θα ψηφιστούν ούτως ή άλλως. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι για να μπορέσει κανείς να έχει μια υπεύθυνη θέση επί του θέματος, χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Ε, βεβαίως είναι δικιά σας ε, η απόφαση και βεβαίως από αυτό το γύρω αργότερα, αλλά θα ήθελα να ξανασκεφτείτε λίγο γιατί πρόκειται για μια πραγματικά δημοκρατική διαδικασία. Πολύ ωραία. Which is uh, of the... Συνεχίζουμε λοιπόν με το σημείο 7 της ημερησίας διατάξεως που προβλέπει έλεγχο των κατεξουσιοδότηση ε, πράξεων και εκτελεστικών μέτρων, μυθή και μυθείο. Έχουμε σημαντικές ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις που έχουν προχωρήσει ε, αρκετά. Θα ε, τις δούμε αυτές, καθώς επίσης και τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα γιατί πρέπει να γίνει και από αυτόν έγκαιρα η συζήτηση πριν ολοκληρωθούν οι κατεξουσιοδότηση πράξεις. Επίσης, δράτω με τις ευκαιρίες για να καλωσορίσω την άτυπη συμφωνία όσον αφορά την νομική ε, αναθεώρηση του προσχεδίου ε, που θα μειώσει από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν σχετικά με τις τεχνικές τροποποιήσεις οι οποίες μπορεί να καθυστερήσουν ε, την ε, ε, περίοδο αντίρρησης από την άλλη πλευρά και αυτό είναι σημαντικό για το Κοινοβούλιο και νομίζω ότι εδώ εκφράζω και αρκετά μέλη του Κοινοβουλίου από καθαρά τεχνική άποψη αυτό είναι ενδιαφέρον και βεβαίως ε, το Κοινοβούλιο δεν θέλει περισσότερα πολιτικά ζητήματα να αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο που μπορεί ενδεχομένως να μειώσει τη διαφάνεια. Ε, κυρίως μεταξύ ΕΣΜΑ και Κομισιόν. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Μάρτιν Μέρλιν, ο οποίος είναι επικεφαλής της ΕΦΙΣΜΑ, καθώς επίσης και τον πρόεδρο της ΕΣΜΑ. Καλωσορίσατε στην ε, Επιτροπή, στην Επιτροπή μας. Και ο κύριος Μέρη και ο κύριος Μέιτζορ θα μας κάνουν ε, μια σύντομη παρέμβαση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα. Έχουμε εγκρίνει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την MIFID 2 το 2014 για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα, την ε, ακαιρεότητα και την ανθεκτικότητα των ε, χρηματοπιστωτικών αγορών. Αυτό θα επιτευχθεί για να, με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθούν περισσότεροι στόχοι όπως είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια, περισσότεροι, περισσότερες συναλλαγές σε τακτικές αγορές και περισσότερος έλεγχος στον τομέα των παραγωγών διευκόλυνση της πρόσβασης σε κεφάλαιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και φυσικά και παρακολούθηση των τεχνολογικών αλλαγών, ιδίως μέσω της ρύθμισης για τις συναλλαγές υψηλής ταχύτητος. Αυτή ήταν η στόχη λοιπόν. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να εφαρμοστούν από την 3η Ιανουαρίου 2017 και αν εξετάσουμε το χώρο των κατεξουσιοδότηση πράξεων, πράξεων λοιπόν οι οποίες δεν βασίζονται στα δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα της ΕΣΜΑ. Υπάρχουν τέσσερις κύριες περιοχές για τις οποίες η, η Κομισιόν, η ΕΣΜΑ, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ομάδος για τις Αγορές Αξιογράφων και οι συγητέ επεξεργάζονται και οι συγητέ επεξεργάζονται. Όλα αυτά θα είναι πολύ σημαντικά για τη σημερινή μα συζήτηση. <clears throat> Πρώτα απ' όλα πρέπει να συμφωνήσουμε για ένα αριθμό ορισμών, σημαντικών ορισμών. Θα πρέπει να θεσπίσουμε κριτήρια και κεφάλαια για εσωτερικές ε, διεργασίες. Ο ορισμός του, της, των συναλλαγών υψηλής ταχύτητας και το τι σημαίνουν παράγωγα και πάνω σε βασικές ε, ποιότητες, βασικές, βασικά αγαθά. Θα πρέπει να καθορίσουμε τους χώρους όπου μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι αγορές. Τρίτον, θα πρέπει να έχουμε τους κανόνες για τη λειτουργία των αγορών που οδηγούν σε ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για την αρχική έκδοση και την μεταγενέστερη έκδοση αξιογράφων και επίσης για τους ε, για τις περιοδικές εκθέσεις που θα πρέπει να δίνουν οι εκδότες αξιογράφων και τέταρτον θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τους κατάλληλους κανόνες στον, στον, ε, σε ό,τι αφορά τα κίνητρα τονίζοντας κάτω από ποιες συνθήκες είναι αποδεκτά, αποδεκτή η παροχή κινήτρων και σε ποιες περιπτώσεις <clears throat> η έρευνα για επενδύσεις δεν αποτελεί από μόνη της ένα κίνητρο και μπορεί να γίνει αποδεκτή από την πλευρά των διαχειριστών χαρτοφυλακίων και των ανεξαρτήτων συμβούλων. Η Κομισιόν δεν έχει καταλήξει σε οριστική άποψη για το πώ θα προχωρήσει για τα θέματα αυτά. Η σημερινή συζήτηση πιστεύω θα διαλευκάνει ορισμένα από αυτά τα θέματα και θα βοηθήσει την απόφαση της Κομισιόν. Σίγουρα όμω είναι κατεπήγον να μπορέσει να υπάρξει μια συνένεση και να προχωρήσουμε ταχαίω ώστε να δώσουμε μεγαλύτερη σαφήνεια και στου συμμετέχοντε στην αγορά και στι εθνικέ αρχέ ε, πριν από την εφαρμογή των νομοθετημάτων αυτών. Αναφέρθηκα στι κατεξουσιοδότηση πράξη. Τώρα έχουμε στα δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα. Εδώ η Κομισιόν παρακολουθεί το έργο τη ΕΣΜΑ, τη Αρχή για τις ε, Αγορές ε, Αξιογράφων. Ξέρετε ότι υπήρξε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τη DG FISMA και τη ΕΣΜΑ για να υπάρξει μια έγκαιρη νομική εξέταση των δεσμευτικών αυτών τεχνικών προτύπων με στόχο να εξασφαλιστεί ότι η ποιότητα της νομικής διατύπωσης ευθυγραμμίζεται με το κοινοτικό κεκτημένο, αλλά φυσικά δεν προκαταλαμβάνουμε με τον τρόπο αυτό το δικαίωμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΜΑ για να καταλήξει σε μια τελική θέση για το σχέδιο δεσμευτικών τεχνικών προτύπων, ούτε προκαταλαμβάνει φυσικά το δικαίωμα της Κομισιόν να τροποποιήσει ή να απορρίψει κάποια από αυτά τα πρότυπα από τη στιγμή που έχει υπάρξει η επίσημη ανακοίνωσή τους προς την Κομισιόν. Παραμένουμε λοιπόν την ακαιρεότητα της διαδικασίας η οποία προβλέπεται από τον κανονισμό της ΕΣΜΑ. Για τα δεσμευτικά λοιπόν <clears throat> τεχνικά πρότυπα, τα κύρια θέματα που μας απασχολούν είναι η διαφάνεια πριν και μετά από μια συναλλαγή στις αγορές, η απουσία ε, προνομιακής μεταχείρισης από τους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους και τις ε, αγορές, αντιμετώπιση της αλγοριθμικής, ε, αλγοριθμικών συναλλαγών και επίσης κατόφλια για να καθοριστούν οι ε, παράπλευρες δραστηριότητες στον τομέα των παραγωγών που συνδέονται με βασικά προϊόντα commodities. Αυτά είναι λοιπόν θέματα στα οποία δίνουμε εμείς την πρέπουσα σημασία. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή και τους ε, σκιοδησηγητές, τον κύριο Φέρμπερ, την κυρία Σουίμπερν, Ντότζ, Βανόιβεν Χόιζεν, Γκίνγκολτ και Ντεμάσι για την πολύ καλή συμβολή τους μέχρι στιγμή στο νομοθέτημα αυτό και πιστεύω ότι είναι κεφαλαιόδες να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο του να εγκριθεί το κείμενο αυτό να, προχω... να υπάρξουν οι εφαρμοστικές διατάξεις στο κείμενο του Ιουνίου 2014 και να έχουμε την απαραίτητη <clears throat> διαφάνεια και σαφήνεια. Είναι πολύ σημαντικό το έργο μας επίσης σε ό,τι αφορά το γενικότερο στόχο πολιτικής του να δημιουργηθεί μια ένωση κεφαλαίου αγορών και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Πρέπει να επιτύχουμε τους στόχους του να τονώσουμε την οικονομική ανάπτυξη να διατηρήσουμε μια αποτελεσματική προστασία των επενδυτών και να προωθήσουμε την χρηματοπιστωτική σταθερεότητα, έχοντας πάντα υπόψη μας το σωρευτικό αποτέλεσμα των διαφόρων νομοθετημάτων που έχουν εγκριθεί και την ανάγκη να αποφύγουμε απρόβλεπτες συνέπειες. <clears throat> Πιστεύουμε ότι η MIFID 2 θα συμβάλλει ιδιαίτερα στην επίτευξη των στόχων αυτών. Για να το πράξει όμως αυτό, θα πρέπει να υπάρξει η σωστή βαθμονόμηση και περάτωση στον τομέα όλων αυτών των μέτρων που ανέφερα. Σε ό,τι αφορά, τη διαδικασία, και κλείνω εδώ κύριε Πρόεδρε, τα δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα θα πρέπει να εγκριθούν μέχρι το Σεπτέμβριο από την ΕΣΜΑ και οι κατεξουσιοδότηση πράξεις θα πρέπει να εγκριθούν από την Κομψιόν και αυτές κατά το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον πρόεδρο της ΕΣΜΑ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε. Αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που με προσκαλέσατε στην ΕΚΟΝ για να παρουσιάσουμε το έργο της ΕΣΜΑ σε ό,τι αφορά το ΜΥΦΙΔ 2 ε, για τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση και θα ήθελα να σας πω ότι ήταν πάντα πολύ επικοδομητική η συνεργασία στις προηγούμενες αιτίε για την σημαντική αυτή νομοθέτηση. Ε, το MIFID 2 και το MIFID είναι το πιο μεγάλο όγκος νομοθεσία σε δεύτερο επίπεδο που έχει πραγματευτεί ποτέ η ΕΣΜΑ. Τώρα κάναμε λοιπόν γύρους ε, διαβουλεύσεων και λάβαμε πολύ καλές και θετικές ε, παρατηρήσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης, περιοδικώς ε, ενημερώνομαι πάνω από το Κοινοβούλιο για τα βασικά στοιχεία των τεχνικών προτύπων και σήμερα θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρεις ε, τομείς, οι οποίοι τονίζονται ιδιαίτερα από τους εμπλεκόμενους φορείς. Η διαφάνεια non-equity, τα παράγωγα πρώτων ύλων και οι χρηματοοικονομικές οντότητες. Δεν θα επισέλθω σε σχόλια για τα τεχνικά, τις τεχνικές συστάσεις, γιατί πλέον τα πράγματα είναι στο γήπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα επικεντρωθώ σε αυτά τα τεχνικά πρότυπα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά το καθεστώς διαφάνειας εκτός μετοχών, θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε τα μερικά συστήματα θα πρέπει να είναι λειτουργικά στην πράξη. Η ΕΣΜΑ έχει αναλύσει ε, μεγάλα, ε, μεγάλο όγκο δεδομένων προκειμένου να βρει συνολικές λύσεις. Δεν θα βρούμε ένα ιδανικό σύστημα που θα ισορροπεί απόλυτα την διαφάνεια με τη ρευστότητα και τα συμφέροντα όλων των συμφερόντων. Όταν ρωτήσαμε στις διαβουλεύσεις ε, ποιο θα ήταν αυτό το σύστημα, το τέλειο σύστημα, ήταν πολύ διαφορετικές οι απαντήσεις. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε ε, εφικτούς συμβιβασμούς και θα κοιτάξουμε τους σχετικούς κανόνες όταν εντοπίσουμε τα βασικά, τις βασικές αδυναμίες. Και αυτό είναι φυσικά το πλεονέκτημα του να υπάρχουν τέτοια τεχνικά πρότυπα προσαρμόσιμα βάσει των εξελίξεων στις αγορές. Να σας διαβεβαιώσω επίσης ότι αναλογιζόμαστε να διαμορφώσουμε ένα πιο ευέλικτο σύστημα το οποίο θα αποτυπώνει πιο καλά τις εξελίξεις στην αγορά και θα έχει πιο καλή βάση δεδομένων και αυτό θα καταστεί πραγματικότητα όταν θα εφαρμοστεί και το MIFIR σε ό,τι αφορά την διαφάνεια το, της αγοράς ε, ομολόγων και το καταβάλουμε προσπάθειες και κατά πάσα πιθανότητα θα διαφέρει το σύστημα από αυτό που διαφάνει στην ε, διαπραγματεύσεις. Τώρα, για να δούμε ποια είναι τα όρια των θέσεών μας, γιατί ακούσαμε πολλές ανησυχίες διαφόρων ειδών. Εξετάζουμε λοιπόν το ζήτημα αυτό και θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη ότι η απαιτήσει για τις θέσεις τέτοιων όριων είναι μεγάλος ε, εύρος ποικιλία από μικρή έως πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα. Και έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε μια λύση που θα ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι η εθνική οι θύνοντες θα πρέπει να θέσουν τις θέσεις ε, ορίων και όλα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν μετά από γνωμοδότηση του, σώματος, του αρμόδιου σώματος της ΕΣΜΑ για να υπάρχει και συνέπεια αλλά και ρευστότητα. Ο τρίτο τομέα, ο οποίο σε πολλέ περιπτώσει αναφέρεται από τους διαβουλευόμενου, είναι το θέμα των ελέγχων. Η ΕΣΜΑ έχει ε, προβλέψει ένα τεστ, ε, έναν έλεγχο πρώτου επίπεδου βάσει των σχεδικών αναλύσεων και πάλι λοιπόν μπορείτε να περιμένετε ένα κείμενο με μεγαλύτερη εξειδικευσή. Εδώ πάλι μας απασχολεί η έλλειψη υψηλής ποιότητας δεδομένων. Είμαστε σίγουροι ότι θα χρειαστεί κι άλλος ένας γύρος ε, ε, προσαρμογή των δεδομένων. Τώρα, επιτρέψτε μου να κάνω κάποια γενικά σχόλια για να τονίσω το εξή ότι πρόκειται για την τεχνική και νομική ποιότητα του κειμένου. Το θέμα ε, δεν είναι να προκαταβάλουμε σε καμία περίπτωση είτε για το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΕΣΜΑ είτε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πώ θα διαμορφώσουν την άποψή του. Κοιτώντα τι διαφορέ που υπάρχουν στι τοποθετήσει, θα πρέπει να σα πω ότι αυτή τη γραμμή θα ακολουθήσουμε και όντως ε, εστιαζόμαστε στην ε, θέματα νομικής ποιότητας για να επιταχύνουμε την όλη διαδικασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος και τώρα να δώσω το λόγο στον εισηγητή, στον κύριο Φέρντερ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τις ε, παρουσιάσεις αυτές από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΕΣΜΑ. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πολύ καλή και στενή συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Φίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία των τελευταίων ετών, γιατί νομίζω ότι ήδη καταφέραμε και πετύχαμε σε κάποια σημεία να βελτιώσουμε σημαντικά τις προτάσεις, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ε, διάφορα ζητήματα στα οποία θα πρέπει να εξκύψουμε. Και θα πρέπει να βελτιώσουμε και να διευκολύνουμε τον τρόπο εργασία μας στα σημεία αυτά. Είναι καλή η συνεργασία με την ΕΣΜΑ, αλλά θα πρέπει να μιλήσουμε και για κάποιες διαδικασίες, για κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τα οποία θα πρέπει να τα επιλύσουμε. Ζητώ κατανόηση, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα. Την, ε, τα positions, limits, τις αγορές ρευστών, ε, ε, την έγκριση προϊόντων και πολλά άλλα. Και νομίζω ότι σε πολλά σημεία Έχουμε ήδη εργαστεί σκληρά, αλλά το γεγονός είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει και θέλει να ε, υποβάλει μόνο δύο μεγάλα πακέτα. Άρα θα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, άλλα νομοθετήματα, στις πράξεις κατά εξουσιοδότηση είναι πιο περιορισμένο το ευρώ και έτσι είναι πιο εύκολη συζήτηση. Να ξεκινήσω από το position limit, από, τις, ε, από τα όρια θέσεων. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το στόχος είναι να εξετάσουμε σύμβαση ανασύμβαση και να ορίσουμε τα όρια ανασύμβαση. Όπως είπατε υπάρχουν αγορές με μεγάλη και πολύ μικρή ρευστότητα στον τομέα αυτό. Και δεδομένου ότι μιλάμε για άνω των χιλίων συμβάσεων και η βάση δεδομένων δεν είναι ιδανική, πρέπει να πω ότι κατανοώ τις πρακτικές δυσκολίες. Η πρόταση δε της ΕΣΜΑ για να εξετάζονται 25% των συμβάσεων με ε, περιθώριο 15 πάνω 15 κάτω ε, δεν είναι σωστό γιατί για τις αγορές με ρευστότητα, με ρευστότητα αυτό το όριο είναι πολύ ψηλό ενώ για αγορές με πολύ μικρή ρευστότητα δεν αρκεί το πόσο αυτό εξετάσαμε τι γίνεται και στις ΕΠΑ. Ορίζονται, προτείνεται να οριστούν μόνο για 28 συμβάσει τέτοια όρια. Αλλά αυτό δεν ε, επαρκεί. Εκεί όμω έχουν και αυτοί το ίδιο πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε το τι θα κάνουμε στο θέμα αυτό. Δεν ε, πιστεύω ότι με την προσέγγιση αυτή θα βγάλουμε άκρη. Το είπατε κι εσείς, ε, ότι δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε μία ενιαία λύση για όλους. Επαναλαμβάνω, αυτό το όριο είναι πολύ υψηλό για τις ρευστές αγορές και πολύ χαμηλό για τις αγορές όπου δεν υπάρχει ρευστότητα. Άρα δεν μπορούμε να το λύσουμε αυτό ε, με μία μόνο λύση. Είναι απαράδεκτο. αυτό. Εξαίρεση της ε, συμπληρωματικής δραστηριότητα. Ε, να υπάρχει άδεια τραπεζική ή να μην υπάρχει. Όποιος ε, δεν εξαιρείται χρειάζεται τέτοια έγκριση, Όποιος εξαιρείται δεν χρειάζεται. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τις άδειε στις τραπεζικές. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προχωρήσουμε με μεγάλη προσοχή για το πώς θα οριστούν οι ωριακές τιμές και χαίρομαι για το ότι η ΕΣΜΑ ανακοίνωσε ότι πρόκειται να ελέγξει το σύνολο του κλάδου. Αλλά και θα κλείσω γιατί αυτό πρέπει να το συζητήσουμε για πολλά θέματα, θα πρέπει να προσέξουμε να μην υπερβάλλουμε συμφωνούσαμε πάντα σε επίπεδο 1 ότι όπου λαμβάνει η χώρα το εμπόριο θα πρέπει να εφαρμόζονται και οι κανόνες για το εμπόριο. Όπου λοιπόν υπάρχει δραστηριότητα χρηματιστηριακή θα πρέπει να τηρούνται και σχετικοί ε, κανόνες για την ε, χρηματιστηριακή λειτουργία και αυτό το ζήτημα με την εξαίρεση για την παραπλαναστριότητα θα πρέπει να ισχύει. 0,5% του μεριδίου της αγοράς. Δεν ξέρω κατά πόσον ε, έχει, είναι σκόπιμο να εφαρμόσουμε αυτό το όριο όπου δεν μπορούμε να ελέγξουμε το κριτήριο της συμμετοχής της αγοράς γιατί δεν έχουμε στοιχεία για την αγορά. Ένα μεγάλο θέμα είναι και η προστασία του καταναλωτή ασφαλώς. Εδώ, συνειδητά και το τονίζω αυτό συνειδητά. Προβλέψαμε μεγάλο περιθώριο για τις εθνικές αρχές. Γιατί, γιατί έχουμε μεγάλο εύρος κανόνων προστασίας του καταναλωτή και πολύ έχουν καταθέσει διάφορες προτάσεις για τις εθνικές αγορές για την εθνική προστασία του καταναλωτή. Και έχουν καταθέσει και νομοσχέδια και πολύ απλά δεν μπορεί, δεν είμαστε σε θέση και είναι και πολιτικά λανθασμένο να βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να πει σε όλο τον κόσμο πώς πρέπει να λειτουργήσει. Αλλά αυτό με τη σειρά του σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η προστασία του καταναλωτή θα πρέπει να διαμορφωθεί όχι με κανονισμό κατά εξουσιοδότηση, αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε τουλάχιστον δύο-τρία έγγραφα για να δώσουμε επαρκέ περιθώριο στους εθνικού νομοθέτες. Διαβουλεύσει. Ε, για τα περιθώρια. Ορίσαμε ότι η ποιότητα για την παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να βελτιωθεί. Άρα, Τα ταχθήκαμε κατά μιας γενικής απαγόρευσης ε, ε, παροχής υπηρεσιών σε ό,τι αφορά το κριτήριο βελτίωση τη ποιότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι και εφικτό. Αν είναι ανέφικτο, ουσιαστικά πάλι θα ισχύει μια απαγόρευση de facto. Και θα πρέπει λοιπόν τα διάφορα μοντέλα να έχουν ένα περιθώριο ε, λειτουργίας, γιατί η Ευρώπη είναι ενωμένη στην ποικιλομορφία της, όχι στην ενότητά της. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να ε, λυθεί λυθεί για το Acton Research, για την έρευνα αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε δύο εθνικές ε, αρχές, οι οποίες καταλήγουν σε διαφορετική α, διαπίστωση και τοποθέτηση. Αυτό σίγουρα θα πρέπει να το συζητήσουμε σε ό,τι αφορά τις ε, υποχρεώσεις δημοσίευσης. Ε, στην ΕΣΜΑ ε, προβλέπεται ένα τέτοιο, μια τέτοια διάταξη για την δημοσίευση των κόστους και των τελών. Υπάρχει, λοιπόν, υπάρχουν και διάφοροι τέτοιοι παρόμοιοι κανόνες και ο στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι για το ίδιο προϊόν ισχύουν στα τρία νομοθετήματα, TRIPS, MIFID και MIFID, ε, οι ίδιες νομικές διατάξεις. Θα πρέπει να ισχύουν λοιπόν τα ίδια για το εκάστοτε προϊόν. Γιατί δεν νομίζω ότι αποτελεί πρόθεση του νομοθέτη κάτι διαφορετικό. Πώς μπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα των διαφορετικών ε, διατάξεων. Στο 26.2 άρθρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποδεικνύει το πρόβλημα αυτό και αναφέρει ότι οι υποχρεώσεις αυτές, ε, αυτές τα διάφορα νομοθετήματα δεν είναι ε, συντονισμένες, δεν είναι εναρμονισμένες. Το επόμενο θέμα Regional Commercial Basis. Στην αρχή προσπαθήσαμε λοιπόν να ορίσουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό και η πρόταση στην παρούσα φάση της ΕΣΜΑ είναι μία σειρά κανόνων για τις διαφάνειας με ένα reasonable margin, με ένα εύλογο περιθώριο. Ουσιαστικά δηλαδή προσπαθούμε να ορίσουμε κάτι το οποίο είναι ασαφές με άλλον έναν όρο που και πάλι είναι ασαφές. Ένα άγνωστο προσπαθούμε να το ορίσουμε με ένα άλλο άγνωστο. Δεν νομίζω ότι μας, μας προχωράει ιδιαίτερα αυτό και μας βοηθάει. Θα ήθελα να καλέσω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει έναν ορισμό που θα εξασφαλίσει ότι υπάρχουν ίσοι κανόνες και δεν θα είναι ελεύθερο προς ε, ερμηνεία ένα δεύτερο σημείο το οποίο πρέπει να σχολιάσουμε με αρνητικό τρόπο, άρθρο 11.2, ότι η αύξηση των τιμών μπορεί να ε, πηγάζει μόνο από αύξηση του κόστους. Νομίζω ότι αυτό είναι υπερβολικά περιοριστικό και θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις επιπρόσθετες υπηρεσίες ενδεχομένω. Ιδάλλως ε, περιορίζουμε την ανάπτυξη. Συστημική εσωτερικοποίηση. Σημαντικό το θέμα αυτό. για τα δίκτυα αυτά και σε ό,τι αφορά την εσωτερικοποίηση των ζητημάτων αυτών. Η ΕΣΜΑ έλαβε την εντολή από τον νομοθέτη στο να ορίσει σε ό,τι αφορά τι τεχνικέ συστάσεις ποια είναι τα κριτήρια για την ε, διαβάθμιση και στον ε, νόμο αντιπέδου 1 προβλέπεται ότι το εμπόριο θα πρέπει να γίνεται συστηματικά και συχνά. Άρα, μπορεί ο αριθμός των ε, φορέων να είναι σταθερός και έτσι να μην υπάρχουν συχνές αλλαγές. Προκειμένου να μιλάμε για συστημική συντορικοποίηση θα πρέπει το συνολικό όγκος για ένα εμπορίο ένας προϊόντος να είναι γνωστός. Αυτό δεν είναι όμως ε, σίγουρο αν ε, μιλάμε για το MIFID 2. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλίσει η ΕΣΜΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όντως διατίθενται τα δεδομένα αυτά για το κριτήριο της ε, ουσιοδούς βάσης, substantial basis, χρειάζομαστε όρια και ένα ελάχιστο κάτω όριο, το όριο για να αποφύγουμε ε, υπερβολική, μάλλον εταιρείε που έχουν χρέους να ε, θεωρούνται ότι εστερκοποιείται το κόστος αυτό. Ένα τελευταίο ζήτημα, όπου έχω δυστυχώς την αίσθηση ότι για ένα σημαντικό ρυθμό αριθμό ζητημάτων στα position limits σε ό,τι αφορά τον ορισμό των waiver του εμπορίου υψηλής συχνότητας και το καθεξής είμαστε λίγο εκτός. Αφενός γιατί η κατάσταση με τα βασικά δεδομένα είναι ασφαλμένη, αφετέρου γιατί τα τεκτενόμενα στην αγορά μετά από την πλήρη εφαρμογή του MIFID κατά πάσα πιθανότητα θα τροποποιηθεί. Άρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο σε διάφορα σημεία να πρέπει να κάνουμε μια εκ των υστέρων προσαρμογή. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να έχουμε και υπόψη μας ποιος θέλουμε να είναι στόχος των κανόνων. Και ανακύπτει λοιπόν το εξή ερώτημα. Τι δυνατότητε υπάρχουν, πόσο γρήγορα μπορούμε να κάνουμε τέτοια προσαρμογή, πώ θα ληφθούν υπόψη και θα εξασφαλιστούν τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερω προ την ΕΣΜΑ μας αναφέρεται συνέχεια ότι μας διαβιβάζονται στις νέες εκδόσεις των κειμένων όταν επιβεβαιώνονται από την ΕΣΜΑ και από το Συμβούλιο της ΕΣΜΑ. Αλλά όταν ε, είναι ολοκληρωμένη η εργασία αυτή δεν μπορούμε να αλλάξουμε πλέον τίποτα. Ζητώ λοιπόν την κατανόησή σας. Θέλουμε κι εμείς ως Κοινοβούλιο να μην αποποιηθούμε των δικαιωμάτων μας. Γι' αυτό λοιπόν θα ήμουν ε, ευγνώμων αν θα μπορούσατε να μου απαντήσετε. Ε, συγγνώμη που μακρηγόρησα και επικεντρώθηκα στα πλέον σημαντικά. Να ζητήσω και συγγνώμη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και να μας πει όμως γιατί μας έδωσε μόνο δύο πράξεις κατά εξουσιοδότηση, ενώ έχει λάβει πάνω από 100 εξουσιοδότησεις. Ευχαριστώ για την ε, πολύ πλούσια και γεμάτη στοιχεία παρουσίασή σας. Thank you. Κυρία Ντότς, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ίσως θυμούνται οι συνάδελφοι ότι την τελευταία φορά που συζητήσαμε για την MIFID 2 και την MIFIR ε, ο κύριος Μάζορ ε, είπε ότι πρόκειται για σημαντικά, ε, ίσως τα σημαντικότερα στοιχεία σε επίπεδου 2 που αντιμετώπισε η ΕΣΜΑ, αλλά τώρα βλέπουμε ότι είναι και από τα πιο ογκώδη νομοθετήματα. Είναι περίπλοκο το θέμα και γι' αυτό θα πρέπει να το δούμε με την δέουσα προσοχή. Ε, θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και την ΕΣΜΑ και την Κομισιόν ε, για την ε, πολύ σημαντική εργασία που έκαναν, γιατί αυτό δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Στην MIFID 2 και, στη MIFID, και στην MIFIR είναι πάρα πολύ σημαντικές και, οι και τα δεσμευτικά τεχνικά πρότυπα, αλλά και η κατεξουσιοδότηση πράξης και επομένως δούλευσαν πάρα πολύ σε αυτό το επίπεδο 2 ε, τους τελευταίους μήνες, όπως άλλωστε και ο εισηγητής και οι εισηγητές. Ελπίζω ότι και η δικιά μας εργασία ε, θα υποβοηθήσει την ΕΣΜΑ και την Κομισιόν ε, Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο καθένας μας μπορεί να μιλήσει για πάρα πολλή ώρα για το κάθε ένα θέμα ε, της ε, ΕΣΜΑ, αλλά νομίζω ότι εγώ θα περιοριστώ στα πιο ε, αμφιλεγόμενα σημεία, τουλάχιστον αυτά που κατά την άποψή μου είναι τα πιο αμφίσιμα και επί των οποίων θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Πρώτα απ' όλα, η προστασία των επενδυτών. Νομίζω ότι ε, όλοι οι εμπλεκόμενοι ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό και βεβαίως ε, κατά μείζωνα λόγο το Κοινοβούλιο. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ε, αυτοί οι οποίοι παρέχουν επενδυτικές συμβουλές το κάνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο χωρίς σύγκρουση συμφερόντων που θα τους απέτρεπε από το να δώσουν τις σωστές ε, ε, ε, πληροφορίες και επομένως συμβουλές στον ενδεχόμενο επι, επενδυτή. Κατά αυτή την έννοια θα πρέπει να αποφευθεί και οποιαδήποτε επιρροή ε, από, ή, παρέμβαση από οποιαδήποτε άλλη ε, εταιρεία. Ε, προβλέπονται μονάχα κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι πολύ προσεκτικά διατυπωμένες. προτείνω μάλιστα να τροποποιηθεί και το σχετικό κεφάλαιο της, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε οι, οι εξαιρέσεις να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες και να αφορούν συγκεκριμένες διαδικασίες. Επίσης, ε, ε, ε, οι διαχειριστές χαρτοφυλακίων θα πρέπει οπωσδήποτε να δεσμεύονται, λέει το κείμενο, από την ποιότητα της εργασίας τους. Ναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποια πιο συγκεκριμένη διατύπωση σχετικά με αυτήν την ποιότητα. Επίσης, ε, μέχρι ποιο βαθμό ε, η επενδυτική προσέγγιση ε, μπορεί να θεωρηθεί ως παρέμβαση. Πιστεύουμε ότι εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία. Ξέρω ότι η ΕΣΜΑ έχει προσπαθήσει να αποσυνδέσει ε, ε, τις πληρωμές ε, από την ποιότητα και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε από την πλευρά του κλάδου. Πιστεύουμε ότι ε, είναι σωστές οι συμβουλές που έχει δώσει η ΕΣΜΑ μέχρι τώρα, ωστόσο ε, κάποιοι ε, ρυθμιστές σε εθνικό επίπεδο ερμηνεύουν διαφορετικά το κείμενο. Ε, ορισμένοι ρυθμιστές θεωρούν ότι ε, ε, κάποιες διαδικασίες είναι επιτρεπτές, άλλοι ότι το κείμενο της Κομισιόν το απαγορεύει. Αλλά δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε περιθώρια για διαφορετικές ερμηνείες σε ένα τόσο σημαντικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα λοιπόν να μας πει η Κομισιόν εάν αυτές οι απαγορεύσεις είναι δεσμευτικές ή όχι. Ο κύριος Φέβρουρ προηγουμένως αναφέρθηκε αναφέρθηκε σε ένα τέτοιο, ε, ε, ε, σε αυτό το θέμα λέγοντας ότι θα πρέπει να έχουμε και ένα περιθώριο ελιγμών, δεν ξέρω αν το εννοούσε πραγματικά. Αυτό που είναι σημαντικό κατά την άποψή μου είναι να αρθεί οποιαδήποτε ανασφάλεια ή αμφιβολία ε, ε, δικαίου. Επίσης τα commodity derivatives είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και για τους σοσιαλιστές ε, αποτελεί προτεραιότητα έτσι ώστε να μην αλλάζει η ε, τιμή ή να μην τροποποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ε, η τιμή βασικών αγαθών, καταναλωτικών αγαθών, ε, είτε είναι τρόφιμα είτε είναι καύσιμα, μέσα από διαδικασίες του, της χρηματαγοράς. Καταλαβαίνω βεβαίως ότι η ΕΣΜΑ θέλει να εισαγάγει κάποια όρια όσον αφορά ε, την ε, ε, αγορά αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί περιέχει πάνω από 1300 στοιχεία, αλλά ε, θα πρέπει να προστατεύσουμε το σωστό τρόπο αυτές κυρίως, αυτούς κυρίως τους τομείς της αγοράς που ε, παρουσιάζουν ιδιαίτερα στοιχεία ρευστότητας. Ε, θα πρέπει να υπάρχει μια βασική γραμμή με την οποία να συμφωνήσει και ο εθνικός ρυθμιστής με παρέκκληση που να μην ξεπερνάει το 15%. Ε, επίσης ε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου σύμφωνα με την παρούσα διατύπωση ένας και μόνο παίκτη ε, μπορεί να έχει το 40% συγκεκριμένη αγοράς. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν και ότι και πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί. Ζητούμε από την ΕΣΜΑ επίσης ε, να ε, ε, επιτρέψει μια πολύ χαμηλότερη θέση που να μην ξεπερνάει το, το 10 έτσι ώστε να επιτρέψει σε, στις συγκεκριμένες αγορές να μην δεσμεύονται από αυτές τις αποφάσεις. Επίσης υπό το άρθρο 57 εδάφιο 3 της ε, ΜΥΦΙΤ ε, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτά τα μη εξαντλητικά 7 ε, στοιχεία τα οποία εκεί αναφέρονται. Κάνουμε συζήτηση για αυτό το 15% για να δούμε κατά πόσον αυτή η προσέγγιση είναι πιο σωστή. Η ΜΥΦΙΤ 2 βεβαίως ε, ε, έχει και ε, περιορισμούς όσον αφορά τα reporting limits και αυτή τη στιγμή η Κομισιόν προτείνει τροποποιήσεις για αγορές με πάνω από 30 συμμετέχοντες, αλλά κατά την άποψή μου είναι πολύ ψηλά τα επίπεδα. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν την Κομισιόν να τα χαμηλώσει. Κάτι άλλο που με ενδιαφέρει είναι η εισαγωγή ε, της ε, νέας, ε, μια νέας διαδικασίας διαφάνειας ε, προσπαθεί να την, ε, την, την προσπάθεια αυτή την έχει ήδη ξεκινήσει η ΕΣΜΑ όσον αφορά δηλαδή την διαφάνεια των χρηματαγορών έτσι ώστε ε, να αποφύγουμε καταστάσεις όπως αυτή πρώτης κρίσεως όπου κανείς δεν ήξερε τι συνέβαινε. Είναι πάρα πολύ σημαντική βεβαίω κατά την έννοια αυτή και η υλοποίηση της MIFID 2 έτσι ώστε να υπάρχει ακόμα περισσότερη παρά λίγο λιγότερη διαφάνεια. Θα πρέπει να είναι η λειτουργία της της αγοράς ε, ανοιχτή και καθαρή έτσι ώστε ε, να είναι σωστή. Αλλά βεβαίως ε, σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιοι traders δεν μπορούν και θα ήταν κακό να δημοσιοποιούν τις θέσεις τους. Γιατί υπάρχουν κάποιες εταιρείε οι οποίες έχουν κάποιες, κάποιους περιορισμούς όσον αφορά την αποκάλυψη στοιχείων. Επομένως, για αυτά τα, για τα ε, χρηματοοικονομικά εργαλεία θα πρέπει να ε, είμαστε προσεκτικοί όταν εφαρμόσουμε τους κανόνες της διαφάνειας. Ε, επίσης, πρέπει να πω ότι δεν έχουμε από τον Δεκέμβριο ήδη του 2014 κάποια ένδειξη από την ΕΣΜΑ σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να προχωρήσει όσον αφορά τη διαφάνεια εκτός στους με εκτός μετοχών. Αυτό είναι αγχωτικό ε, και ε, ξέρουμε ότι γίνεται πολλή συζήτηση όσον αφορά τον καθορισμό αυτών των κατοφλίων, αλλά από την ίδια την ΕΣΜΑ δεν έχουμε ακούσει και πολλά. Και νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι σωστό ε, ότι αυτοί οι ίδιοι βουλευτές οι οποίοι ε, έχουν ε, πάρει αποφάσεις και έχουν καθορίσει πληροφορίες όσον αφορά τη διαφάνεια να μαθαίνουν διάφορα πράγματα από δεύτερο χέρι. Και δεν είναι δυνατόν εκ των υστέρων και για περιπτώσεις όπως το RTS να ε, μας υποβάλλονται εκ των υστέρων λέω κάποιες ε, ε, θέσεις για τις οποίες δεν θα μπορέσουμε να έχουμε συζητήσει. Άλλο θέμα, αυτό το Systematic Internalizer. Κοιτάξτε, ναι, θα προσπαθήσω να τα πω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αργήσαμε και λίγο να ξεκινήσουμε, παρότι είμαστε όλοι εδώ. Εν πάση περιπτώσει, Επ' αυτού να πω πολύ σύντομα ότι με απασχολεί λίγο το θέμα. Θα ήθελα η Κομισιόν να ε, πει ε, σαφώς ότι πρόκειται ε, για ένα διμερές εργαλείο μονάχα και επομένως δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται πάντοτε. Επίσης, σε κάθε bilateral trading θα πρέπει η Κομισιόν ε, να ε, ε, καθορίσει ότι οι συνθήκες θα πρέπει να είναι καθαρές και τίποτα να μην γίνεται χωρίς διαφάνεια. Εμείς επίσης θέλουμε να ζητήσουμε να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα είναι αρκετά ευέλικτο διότι αλλάζουν οι τεχνολογίες και παρασύρουν και τροποποιούν και τις ε, την αντιμετώπιση των αγορών καθώς επίσης και τη συμπεριφορά. Ε, και θέλουμε η ΕΣΜΑ να ε, τροποποιείται σύμφωνα με αυτές τις αλλαγές και προσαρμογές. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Να σας υπενθυμίσω ότι δεν έχουμε άπειρο χρόνο, θα πρέπει να δώσουμε την δυνατότητα στην Κομισιόν να απαντήσει. Η ΚΕΙΤ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι τον πιο σύντομη μετά από τις δύο προηγούμενες ομιλίες, αλλά ξέρετε ότι είναι πολύπλοκο το θέμα και είναι δύσκολο να είναι κανείς πολύ σύντομος. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε τώρα ε, είναι να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει ο απαραίτητος έλεγχος και γι' αυτό θα καλύψω και την ε, πρόταση της ΕΣΜΑ και την κατεξιοδότηση πράξη της Κομισιόν. Χρειάζεται να υπάρξει ένα σύστημα ελέγχου γιατί οι αγορές μας δεν είναι τόσο βαθιές και ρευστές όσο οι παγκόσμιες αγορές. Πρέπει λοιπόν το σύνολο αυτών των κανόνων πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως ένα εργαλείο για να βελτιώσουμε το βάθος και τη ρευστότητα στις αγορές μας, να τις κάνουμε πιο ε, ίσες σε επίπεδο ανταγωνισμού και όχι να σταματήσουμε όλες τις ε, συναλλαγές επειδή δεν έχουμε κάνει την σωστή ρυθμίση. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω και την Κομισιόν και την ΕΣΜΑ για την ε, παρουσία τους. Νιώθω ότι κάπως έχουν αλλάξει τα πράγματα και δεν παίρνουμε τις ίδιες πληροφορίες που παίρναμε μέχρι πριν από λίγους μήνες, ιδίως σε σχέση με το RTF. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για το ανοιχτό της πνεύμα και τη θέλησή της να συζητήσει για τις κατεξουσιοδόσεις πράξεις και επίσης το να έχουμε νέες ε, μορφές του, της πρότασης έχει βοηθήσει εμένα και τους συναδέλφους μου να καταλαβαίνουμε το πώς εξελίσσεται η σκέψη σας και ποια προβλήματα αντιμετωπίζετε. Επειδή παίρνουμε πολύ στα σοβαρά την ε, υποχρέωσή μας να ελέγξουμε αυτά τα θέματα, πρέπει να πω ότι έχω κάποια προβλήματα ακόμα με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις και πρέπει να σας πω ότι ένα από αυτά τα θέματα δεν έγινε δεκτό το επιχείρημά μου στον τριγωνικό διάλογο η άλλη πλευρά επέτυχε την δική της, να επικρατήσει τη δική της άποψη. Αυτό είναι λεγόμενη έρευνα των επενδύσεων. Αναφέρθηκε προηγουμένως αυτό και εμείς έχουμε διαφορετικές θέσεις στην Επιτροπή μας. Αυτό είναι και κάτι που να οδηγήσει σε πολιτική συμβιβαστική λύση. Δεν πετυχαίνουμε πάντα ό,τι θέλουμε. Εγώ ποτέ δεν θεώρησα στις συζητήσεις του τριγωνικού διαλόγου ότι είχαμε απαγορεύσει απόλυτα κάθε μορφή επενδυτικής έρευνας που να έχει το χαρακτήρα κινήτρου. Μέσα στο ε, τριγωνικό αυτό διάλογο δεν έχει δεκτή δική μου άποψη, γι' αυτό υποστηρίζω τον κύριο Φέρμπερ, ο οποίος είπε ότι δεν είχαν συμπεριληφθεί οι, τα κίνητρα στην επενδυτική έρευνα και φυσικά αυτό ίσως ήταν ένα ελάχιστο θέμα. Αν συγκρίνεται το κόστος της ε, έρευνας στο συνολικό ύψος των χαρτοφυλακίων και του κόστους διαχείρισής τους, είναι πράγματι περιορισμένη περιορισμένο το κόστος. Πολλές έρευνες που γίνονται δεν οδηγούν ποτέ σε μία <clears throat> συναλλαγή, οπότε γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία εάν δεν αλλάζει την, ε, το ύψος του ενεργητικού που είναι υποδιαχείριση. Νομίζω λοιπόν ότι η έννοια του ελάσσονος θα πρέπει να τροποποιηθεί. Η Κομισιόν θα πρέπει να αντιμετωπίσει λοιπόν το θέμα της έρευνας ε, επενδύσεων ως τμήμα της ε, κεφαλαιοχικής της, αγοράς, της Ένωσης Αγορών Κεφαλαίων. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε περισσότερη ανεξάρτητη έρευνα στην Ευρώπη, πρέπει να ενθαρρύνουμε περισσότερους φορείς να ερευνούν τις επενδύσεις των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών, θα πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα αυτό προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αλλά να το, απο... <clears throat> να το απαγορεύσουμε βάσει τη MIFID 2 δεν είναι κάτι το οποίο είναι πρόσφορο. Η Ένωση Κεφαλουχικών Αγορών είναι μια ευκαιρία να έχουμε μια θετική προσέγγιση και όχι μόνο μια απαγορεύση που δεν θα έχει θετικά αποτελέσματα για τους επενδυτές. Το δεύτερο είναι η λεγόμενη λογική εμπορική βάση. Το 2010 που εργαζόμουν σε μια αντίστοιχη έκθεση, αυτό το οποίο μου λέγανε όλοι είναι ότι είναι πάρα πολύ ψηλό το κόστος των δεδομένων στην Ευρώπη και δεν υπάρχουν εδρεωμένα στοιχεία. <clears throat> αυτό το οποίο ελπίζαμε όταν φτάσαμε στο τελικό κείμενο για τη ΜΥΦΙΤ είναι ότι θα υπήρχε μια λύση και ένας ορισμός του τι είναι μια λογική εμπορική βάση. Νομίζω ότι η πρόταση της Κομισιόν συνδέονται τα τέλη με το κόστος παροχής δεδομένων και με κάποιο λογικό κέρδος για προστιθέμενη αξία, το οποίο θα έπρεπε να αναφέρεται και να δημοσιοποιείται, αυτό θα μπορούσε να συνάδει με την εντολή ε, επίπεδου 1, ώστε να γνωρίσουν όλοι τι πρέπει να πληρώνουν για αυτές τις υπηρεσίες. Αλλά τώρα αναφέρεται ότι πρέπει να είναι η μεθοδολογία που δημοσιοποιείται και όχι το κόστος. Εάν κάποιος θεωρείται είναι προς το οικονομικό του συμφέρον, μπορεί τώρα να μην αποκαλύπτει το κόστος. Αυτό όμως μπορεί να ανατρέψει το όλο σύστημα. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την Κομισιόν να μην είναι κενό περιεχομένου το κείμενό της στο θέμα αυτό. Και έρχομαι τώρα το τμήμα της ε, πρότασης ΕΣΜΑ και θα παραμείνω μονάχα στον τομέα των αγορών. Ξέρετε ότι εγώ νοιάζομαι πάρα πολύ για τις αγορές. Αλλά πραγματικά απογοητεύομαι από τη σειρά των μη εγγράφων, των μη επισήμων εγγράφων που έχει παρουσιάσει ΕΣΜΑ στο Κοινοβούλιο. Πέρα από τη νέα μορφή νομικού ελέγχου, η ΕΣΜΑ θέλει να εισαγάγει διαφάνεια στις αγορές, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνται αυτοί οι κανόνες είναι κάθε άλλο παραδιαφανής, τουλάχιστον για εμάς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σε σχέση με το θέμα του RTF είναι το καθεστώς διαφάνειας πριν και μετά μια συναλλαγή, ιδίω για την αγορά ε, ομολόγων. Θεωρήθηκε ότι αυτό το έγγραφο θα μπορούσε να είναι ένα θετικό στοιχείο στο Ηνωμένο, στις Ηνωμένες Πολιτείες η διάταξη αυτή ξεκίνησε με τις πιο ε, ρευστές κατηγορίες ομολόγων και σιγά σιγά επεξετάθηκε στις υπόλοιπες. Εμείς θα πρέπει και εμείς να ξεκινήσουμε με μια απόλυτα συντηρητική αντιμετώπιση και σιγά σιγά να κάνουμε τους κανόνες μας πιο αυστηρούς και όχι από την αρχή να έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση για όλες τις ε, συναλλαγές και ούτως ή άλλως η διαφάνεια μπορεί να εξεταστεί κυρίως μόνο μετά από μια συναλλαγή και όχι πριν από μια συναλλαγή. Μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα λοιπόν για τα θέματα με τα στοιχεία που έχουμε. Μας είπα η ΕΣΜΟ ότι προσπαθούν να επιλύσουν τα προβλήματα αυτά, αλλά δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω αυτή τη στιγμή κατά πόσο η πρότασή σας, η προσαρμογή που προτείνετε, θα είναι αναλογική και λεπτομεριακή επαρκώς και δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να καλυφθούν όλα αυτά τα στοιχεία που με απασχολούν στη νέα πρόταση. Ελπίζω ότι βελτιώνετε την πρότασή σας όσο περνάει ο χρόνος, λαμβάνετε υπόψη όλα αυτά τα προβλήματα τα ανακύπτουν. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι δεν είναι ίδιε όλες οι αγορές ομολόγων. Δεν μπορεί να υπάρχει μια ενιαία κατηγορία εργαλείων που να είναι κατάλληλη για όλα τα κρατικά ομόλογα, παραδείγματο χάρη. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο θα ήθελα να εξασφαλίσω ότι καλύπτουμε είναι ότι δεν πρέπει να καλύπτουμε, δεν πρέπει να περιλαμβάνουμε στην ανάλυση τις συναλλαγές κάτω από 100.000 ευρώ. Και τέλος θέλω να τονίσω ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια <clears throat> για αυτήν την ε, αντιμετώπιση για να λάβουμε υπόψη και την χρονική στιγμή και όχι μονάχα την βαθμολόγηση των SSTIs. Και αν λάβουμε υπόψη λοιπόν το γεγονό ότι η ΕΣΜΑ θεωρεί ότι η έλλειψη δεδομένων είναι ένα πρόβλημα για τη διατύπωση των κανόνων αυτών, ελπίζω ότι θα είναι έτοιμοι να δεχτούν μια διαφορετική προσέγγιση, να παρουσιάσουν διαφορετικέ επιλογέ, ότι οι χρηματοπιστωτικοί φορεί που έχουν περισσότερα δεδομένα και περισσότερο προπολογισμό μπορούν να του βοηθήσουν να καταλήξουν στου κατάλληλου κανόνε. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο υπακούει στα συμφέροντά τους αν έχετε τη δυνατότητα όλοι αυτοί να χρησιμοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη τους για τα θέματα αυτά. Λόγω των προβλημάτων που έχουμε με τα έγγραφα της ΕΣΜΑ, εγώ φοβάμαι ότι το αυτό το οποίο θα προκύψει μετά από το νομικό έλεγχο και όταν έρθει σε εμά μπορεί να εξακολουθεί να έχει τα προβλήματα αυτά που ανέφερα και δεν έχει πολλές δυνατότητες πια το Κοινοβούλιο για να εγκρίνει ένα τέτοιο έγγραφο οι αγορές μας για τα κρατικά ομόλογα δεν πρέπει να επηρεαστούν αρνητικά λοιπόν από αυτή την έλλειψη επιτυχίας στο εγγραφή της ΕΣΜΑ. Thank you. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κόρα των Ιουέζεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω όπως όλοι οι υπόλοιποι ευχαριστώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΣΜΑ, τον Μάρκους Φέμπε, τον εισηγητή μας και φυσικά όλους τους συναδέλφους για την καλή δουλειά που έχει γίνει ως τώρα. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμα φτάσει στο τελικό μας στόχο και εγώ έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Και ως συνήθως ο διάολος ε, κρύβεται στις λεπτομέρειες και όταν μιλάμε για ορισμούς και τέτοια ζητήματα ε, εξίσωσης, εδώ έχουμε πολλά ερωτήματα. Και να ζητήσω από τους συναδέλφους να διευκρινίσουν κάποια ζητήματα για να δούμε πού βρισκόμαστε για την Γενική Διεύθυνση Υφίσμα τώρα. Κάποια ερωτήματα για την αποκάλυψη, τη δημοσίευση του κόστους. Και ο Μάρκος Πέμπερτ θα έθεσε το ζήτημα αυτό. Καλώ ορίζουμε την ε, ε, αναλογικότητα του άρθρου 56 σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των όρων ε, και των διατάξεων δημοσίευσης Στο 56.2 του κανονισμού για το MIFID η εντολή αναφέρεται στις επενδυτικές ε, εταιρείε που έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν τέτοιες πληροφορίες στους επενδυτές τους, όπου δεν δημοσιεύονται παρκώς αυτές οι πληροφορίες για το κόστος συναλλαγής, για παράδειγμα. Υποχρεώνονται οι εταιρείε αυτές να ε, ε, αξιολογούν, να υπολογίζουν το κόστος αυτό ανταυτού. Θεωρούμε ότι αυτό είναι υπερβολικό και όπως αναφέρεται στις ιδεολογικές σκέψεις θα πρέπει το κόστος αυτό να θεωρείται επαρκές. Ζητούμε δηλαδή από τις εταιρείε να διορθώσουν τα προβλήματα διαφάνειας της εταιρεία παραγωγής των προϊόντων. Αυτό θεωρούμε ότι είναι υπερβολικό. Θα ζητούσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βρει άλλους τρόπους για να διαβεβαιωθεί ότι όλο το κόστος ε, αποκαλύπτεται στον, και δημοσιεύεται στον ε, καταναλωτή. Στο επόμενο ζήτημα, σε ό,τι αφορά τον καθορισμό της αυτοδότητας. Υπάρχει η προσέγγιση εργαλείο-ανεργαλείο και ε, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η προσέγγιση κατηγορίας εργαλείων. Η ΕΣΜΑ σε ό,τι αφορά τα σταθερά εισοδήματα βασίζεται πιο πολύ στην μέθοδο κατηγοριών ε, με συγκεκριμένα όρια σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την ημερομηνία έκδοσης και κάποιες εθνικές αρχές προτιμούν την ανάλυση εργαλείο-εργαλείο μέσα στην κατηγορία εργαλείων. Αυτή η προσέγγιση εργαλείο θα μπορέσει με καλύτερο τρόπο να αντικατοπτρήσει τις ιδιαιτερότητες των μεμονωμένων ομολόγων. Και θα ήθελα να σας ζητήσω ποια είναι η δική σας άποψη για την προσέγγιση εργαλείο ανά εργαλείο και η αναθεώρηση της μεθόδου αυτή θεωρούμε ότι θα βελτίωνε σημαντικά την ακρίβεια για τα α, λανθασμένα στοιχεία, θετικά ή αρνητικά. Δεύτερη ερώτηση. Έχω διάφορες ερωτήσεις βέβαια για το θέμα της ρευστότητα και για τις απαλλαγές για τα πακέτα. Στην προσέγγιση COFI τα πακέτα προϊόντων θα πρέπει να θεωρούνται ε, τα πακέτα εργαλείων θα πρέπει να θεωρούνται διαφορετικά εργαλεία προκειμένου να μην είναι ε, κακή η τιμολόγηση των προϊόντων. Η ΕΣΜΑ πιστεύει ότι έχει εντολή σε επίπεδο 1 για να οριστούν τα πακέτα ως ξεχωριστή κατηγορία εργαλείων σε ό,τι αφορά και απαλλαγές πριν από την εμπορία. Αν ναι, να μας πει η ΕΣΜΑ ποια είναι η άποψή της σε ό,τι αφορά την ε, διαταξή τρέιντων βένιου για τη διαφάνεια, ιδιαίτερα όταν ε, δεν γίνεται η εμπορία των προϊόντων στην ίδια τοποθεσία. Δεύτερον, το πακέτο θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν είναι ρευστό όταν ένα στοιχείο δεν είναι ρευστό ή όταν η πλειοψηφία, η πλειονότητα των ε, αυτών δεν είναι ρευστή. Θα πρέπει να υπάρχει το όριο για αν ένα πακέτο αποτελείται από έναν χειρισμό συστατικών και τρίτον, ο καθορισμός ε, των απαλλαγών πριν από την εμπορία. Θα πρέπει να βρείτε αυτή η απαλλαγή όταν ένα τέτοιο τμήμα ε, ε, δικαιούται απαλλαγή ή μόνο όταν η πλειονότητα δικαιούται απαλλαγή. Και κατά τέταρτον το πακέτο θα πρέπει να κοιτάμε κατά πόσον φτάνει ένα όριο ή θα πρέπει να κοιτάμε την πλειονότητα των στοιχείων του πακέτου. Τελευταία ερώτηση την οποία την έχει θέσει και με λίγο διαφορετική μορφή, νομίζω, η συνάδελφος Αναλής Ντότς, για το καθεστώς απαλλαγής πριν από την εμπορία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αποφευθούν οι παραλλαγικοί κίνδυνοι στην αγορά. Και πολλοί είπαν ότι τα όρια των SSTI και θα πρέπει να μειωθούν. Κάποιοι είπαν ότι θα πρέπει να μειωθεί στο 50%. Πιστεύει η, η ΕΣΜΑ ότι χρειάζεται αυτή η μείωση. Πιστεύω ότι η μια έγκαιρη και πριετική αναθεώρηση των όριων είναι απαραίτητη για να υπάρχει μια σωστή βαθμονόμηση. Ζώτησε ο κύριος Φέρμπερ πόσο γρήγορα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά θα πρέπει να προσέξουμε, να μην προκαλέσουμε ε, ζημιά. Μπορεί να γίνεται λοιπόν εκ νέου βαθμονόμηση κάθε 6 μήνε μέχρι να γίνει αναθεώρηση του συνολικού πακέτου. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα ήταν ε, πολύ σωστό γιατί γίνεται πάρα πολύ μεγάλη η συζήτηση για τα όρια. Γιατί πιστεύει η ΕΣΜΑ για να συμπεριληφθούν ε, εμπορίες κάτω από τα 1000 ευρώ. Ιδιαίτερω ε, επειδή αυτά τα συστήματα εμπορία, αυτέ οι συναλλαγέ είναι συνήθω πολύ πιο μικρέ στον όγκο του από ότι ο μέσος όρος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Επόμενος, ο μιλητής ο Φάμπι Δεμάνσε. I try to be Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο ε, σύντομος. Ευχαριστώ πολύ την ΕΣΜΕ, ευχαριστώ τον εισηγητή, ε, ευχαριστώ και τους ε, σκιώδεις που δούλεψαν σκληρά και έχουν και γνώση του θέματος. Θα πω μόνο μερικά στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την πραγματική οικονομία, τα position limits πρώτα απ' όλα. Ε, ε, η ΕΣΜΑ ζητάει κατά, ε, κατά περίπτωση περιορισμού της τάξης του 40%. Αυτό όμως δεν εμφυγραμμίζεται με τον σκοπό του επίπεδου 1 και είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε γιατί θα πρέπει οι traders να ε, ε, ε, μπορούν να προχωρήσουν σε πάνω από ένα τρίτο των, των ευστοποιήσεων όσον αφορά τα αναλώσιμα. Επίσης πιστεύουμε ότι με αυτή την έννοια θα έχει μεγαλύτερη διακύμανση, volatility η αγορά σε ορισμένες σε περιπτώσεις, ακραίες περιπτώσεις, ε, ε, μπορούμε να δώσουμε κάποιες, να μπορούν να δοθούν κάποιες ε, εξαιρέσεις από τον εθνικό ρυθμιστή χωρίς να γενικεύσουμε την δυνατότητα αυτή. Ε, επίσης πιστεύουμε ότι ε, ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε προς άλλη κατεύθυνση όσον αφορά αυτήν την βασική γραμμή προστασίας. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει προς τα κάτω να ξαναδεί η ΕΣΜΑ τα, τα ε, ε, όρια τα οποία έχει, τουλάχιστον για ορισμένους βασικούς τομείς της ε, αγοράς. Ε, επίσης θα πρέπει να δούμε ποια είναι και η άποψη της ΕΣΜΑ και της Κομισιόν γι' αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά την position reporting, πιστεύουμε ότι θα πρέπει και εδώ από το 30 να φτάσουμε στο 20 ή ακόμα και στο 10, δηλαδή να γίνει αναθεώρηση προς τα κάτω. Η Κομισιόν βεβαίως διατείνεται ότι το 30 είναι πολύ καλύτερο. Υπάρχει όμως το άρθρο 28 ε, άρθρο 28 της ε, πράξης που λέει ότι οι θέσεις ε, δεν είναι απαραίτητο να δημοσιοποιούνται και ότι εν πάση περιπτώσει αγορές δεν παίζει μεγάλη ρόλο, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά εάν το reporting ξεκινάει στο 30 ή στο 20 αλλά σε ορισμένες συναλλαγές ε, τουλάχιστον για, ε, για τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν λιγότεροι από 20 ε, traders, ε, τότε πραγματικά μπορεί ε, αυτό το reporting limit να κάνει μεγάλη διαφορά. Ευχαριστώ, Σβέν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την Κομισιόν και την Έτσιμα για το πολύπλοκο και δύσκολο αυτό έργο του τα περισσότερα θέματα έχουν αναφερθεί από τους συναδέλφους, δεν πρόκειται να τα επαναλάβω. Αλλά θα ήθελα να σταθώ στην προστασία των επενδυτών. Πιστεύουμε ότι οι κανόνες ε, δημοσίευσης, οι οποίοι αναφέρονται από την ΕΣΜΑ, νομίζω ότι καλύπτουν αυτό το κείμενο και αυτά τα οποία έχουμε ψηφίσει θα ήθελα να πω στους συναδέλφους και κυρίως στην Κέιτ ότι δεν υπάρχει καμιά πρόταση να απαγορεύσουμε τίποτα ιδίω σε ό,τι αφορά την ε, έρευνα. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει κανείς με κάλυψη κάποιας άλλης δραστηριότητος. Αν θέλει κανείς να το κάνει όμως πρέπει να το ζητήσει χωριστά και να το πληρώσει χωριστά και θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι ότι είναι μια, κατά κάποιο τρόπο ένα κίνητρο για την επένδυση. Αυτό το οποίο προτείναμε λοιπόν να εφαρμόσουμε στο άρθρο 47 του σχεδίου είναι ίσως κάπως ε, αμφίβολο κατά πόσο καλύπτεται στο επίπεδο 1 για τα θέματα των ορίων θέση θέλω να υπογραμμίσω αυτά που είπε ο εισηγητής και άλλοι ομιλητές. Ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για μένα είναι το θέμα της ερμηνείας που δίδεται στο ίδιο αυτό έγγραφο στο κείμενο. Γιατί αυτή η ερμηνεία τελικά θα οδηγήσει τελικά σε μια επανεθνικοποίηση του καθεστώτος αυτού και μόνο ένα έλεγχο εκ των υστέρων από την ΕΣΜΑ. Το κατά πώς θα λειτουργήσει αυτό είναι αμφίβολο για μένα και νομίζω ότι η ερμηνεία της ε, διατύπωσης το ίδιο το, το ίδιο συμβόλαιο έρχεται σε σύγκρουση με την αιτιολογική σκέψη 131 της ΜΥΦΙΤ και επίσης έρχεται σε σύγκρουση και με άλλα σημεία στην οδηγία όπου αναφέρεται σαφώς ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει παράκαμψη, ότι η ερμηνεία της έννοιας το ίδιο, η ίδια σύμβαση θα πρέπει να σημαίνει ότι είναι το ίδιο έγγραφο σύμβολα, ότι έχει το ίδιο περιεχόμενο. Εν τέλει λοιπόν ο κίνδυνος είναι ότι όλο το σύστημα για, του, για τα όρια θέσεις είναι ότι ορισμένα συμβόλαια τα οποία δεν είναι αρκετά ρευστά για να την χάνουν ρύθμιση και καταλαβαίνω εδώ πέρα αυτά τα οποία είπαν και άλλοι συνάδελφοι φοβάμαι ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε μια κατάσταση όπου τα συμβόλαια για βασικά προϊόντα τα οποία έχουν επαρκή ρευστότητα δεν θα καλύπτονται και η κατεύθυνση που δίδεται από τα πρότυπα δεν οδηγεί σε μια σαφή εγγύηση ότι θα τύχουν τις ε, ρύθμισεις που εμείς έχουμε υποσχεθεί στους εκλογείς μας μετά από την ε, έγκριση της ΜΥΦΙΤ. Το πνεύμα λοιπόν και η ουσία των προτινομένων προτύπων και της κατεξουσιοδότησης πράξης δεν καταδεικνύει ότι ο στόχος τον οποίο εμείς είχαμε συλλογικά θεσπίσει και υπερψηφίσει πράγματι μπορεί να επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο. Τίθεται λοιπόν σε κίνδυνο η αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και στις ίδιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σύνολο σε ό,τι αφορά την ικανότητα να επιτύχει το στόχο της ε, ρύθμισης υπερβολικών και ερδοσκοπικών δραστηριοτήτων που μπορούν να διαταράξουν την αγορά για ορισμένες από αυτές τις ευαίσθητες αγορές βασικών προϊόντων. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να σας ζητήσω να βελτιώσετε τα, τη διατύπωση για τα θέματα αυτά και πρέπει να καταγράψω ότι από διάφορες ομάδες και, τα, και τον ίδιο τον εισηγητή έχουν αναφερθεί αυτά τα προβλήματα, αλλά εσείς δεν έχετε κουνηθεί ρούπι σε σχέση με τα θέματα αυτά. Επομένως, θα πρέπει να λάβετε υπόψη αυτά τα οποία έχει πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι δεν είναι εύκολο το έργο σας. Έχετε ένα διοικητικό, ένα εποπτικό συμβούλιο, μετά έχετε ένα ε, έχετε και την Κομισιόν μαζί σας και μετά έχετε αυτό το ανώτερο του Κοινοβούλιο και σας ζητάει να κάνετε αλλαγές. Αυτό είναι δύσκολο για σας, αλλά αυτό θέλατε να κάνετε και αυτό είναι το έργο σας. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο αριθμό των σχολείων που έχετε ακούσει και τονίζουν ότι τίθεται σε κίνδυνο η πρότασή σας και δεν θα γίνει αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και η πρότασή σας θα πρέπει κάπου να έχει μια αιτιολόγηση του γιατί δεν δεχτήκατε καμία αλλαγή. Αυτή, αν αυτή η προσέγγιση σας να μην αλλάξετε τίποτα, Σα το λέω σαφώ ότι αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι καμία από τι πολιτικέ ομάδε και ευαισθησίε που υπάρχουν και αντανακλώνται στι συμβαστικέ μας λύσει θα αποδεχτούν μια τέτοια απάντηση για όλα αυτά τα θέματα από την ΕΣΜΑ. Και τέλο να υπογραμμίσω ένα σημείο το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ. Όλα αυτά τα οποία κάνουμε εδώ πέρα για την προστασία των επενδυτών στην ΜΥΦΙΤ αυτή τη στιγμή βρίσκονται εν αμφιβόλω σε κίνδυνο γιατί οι διαδικασίες, οι διαπραγματεύσεις του IND2, οι οποίες περατούνται τώρα, μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα ότι μπορεί κανείς να βάλει τα προϊόντα του σε ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο και έτσι όλο το θαυμάσιο έργο σας σε επίπεδο 2 θα ξεπεραστεί γιατί δεν προβλέπεται εκεί επίπεδο 2. Και επίσης σε θέματα δημοσίευση στο καθεστώς MIFID 2 είναι πολύ πιο περιορισμένο. Ζητώ από την Κομισιόν να λάβει υπόψη αυτά τα οποία βρήκαν οι τρει ε, εξειδικευμένοι φορείς. Ξέρω ότι επειδή κουνάτε θετικά το κεφάλι σας, ξέρετε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να το παρακάμψει κανείς με την IMD, αλλά η Κομισιόν δεν έχει κάνει τίποτα για το IMD 2 δεν βλέπω να υποστηρίζετε τη νομική υποστήριξη να υπάρχουν ισοδύναμοι κανόνε για τα προϊόντα που καλύπτονται από την MIFID και τη MIFID 2. Η Κομισιόν ξέρει μονάχα μία φωνή η οποία πρέπει να την εγκαλέσει είναι οι συνθήκες. Ζητώ από την Κομισιόν λοιπόν να υποστηρίξει και να προστατεύσει αυτά που έχουμε συμφωνήσει και στις διαπραγματεύσεις IMD2 και πρέπει να πω ότι όλες οι συζητήσεις εδώ για την προστασία των επενδυτών ακυρώνονται αν μπορείτε απλώς να αλλάξετε το σχεδιασμό του προϊόντος και δεν υπόκειται σε κανόνες δημοσίευσης ή επίπεδου 2 και ουσιαστικά αυταπατώμεθα σε αυτή την περίπτωση θα ήθελα να καταλάβω από την πλευρά της Κομισιόν γιατί δεν τηρεί την νομοθεσία και δεν προασπίζει τις συνθήκες. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά ζητήματα πολιτικά έχουν τεθεί ως ερωτήματα προς εσάς και όντως φαίνεται ότι η ανησυχία για το ζήτημα των παραγόγων πρώτων υλών είναι ένα θέμα που προκαλεί ανησυχίε γενικότερα και φυσικά θα θέλαμε να ακούσουμε με σαφήνεια ποια είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα αυτό γιατί ακούσαμε και σαφή ζητήματα τα οποία έθεσαν οι ομιλητέ, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Να ζητήσω κι εγώ διευκρίνηση για το θέμα της ε, απαγόρευσης ή μη απαγόρευσης CSA. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι το θέμα απαγόρευσης, αλλά ασφαλώς θα ήθελα να μας πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ερμηνεύει το ζήτημα. Και θα ήθελα να, προσθέσω και ένα άλλο σημείο το οποίο δεν ε, το θέσαμε ιδιαίτερος για το... τις ανησυχίες για την αντίκτυπο, αντίκτυπο των συναλλαγών υψηλής συχνότητας για την αγορά κρατικών ε, εθνικού χρέους. Κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι θα πρέπει να μπουν δικλείδε ασφαλεία προκειμένου να αποτραπούν ενδεχόμενε ανεπιθύμητε παρενέργειε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ΕΣΜΕ έχουν το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τα βασικά ζητήματα τα οποία ακούσαμε από τον εισηγητή και από τους κοιόδες εισηγητές. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω, γιατί για μας είναι βασικό να οριστικοποιήσουμε πλέον το κείμενο και να ακούσουμε τις παρατηρήσεις. Για να περάσουμε στα πιο συγκεκριμένα ζητήματα τώρα, να πω για την πλευρά της προστασίας των επενδυτών. ιδιαίτερα για το θέμα αυτό του πώς ε, αντιμετωπίζουμε την έρευνα, θα ήθελα να πω το εξή ότι το κείμενο επίπεδο 1 α, δεν επιτρέπει τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τα κίνητρα για τους διαχειριστές των χαρτοφυλακίων. Αυτό θα πρέπει να γίνει σεβαστό στο επίπεδο 2 και στην εφαρμογή του επίπεδου 1. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να οριστεί το τι αποτελεί inducement, κίνητρο, απαλλαγή, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η απαγόρευση τέτοιων κινήτρων εφαρμόζεται. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΣΜΑ η τεχνική της σύσταση ΕΣΜΑ είναι να εισαχθεί ένας μηχανισμός που θα εξετάζει το πώς θα πληρώνεται, πώς θα αντιμετωπιστεί η έρευνα για να μην θεωρηθεί κίνητρο. Και αυτός είναι ο στόχος των όσων συζητούσαμε μαζί σας και με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες στο EZSE. Να διευκρινίσω επίσης ότι από το 2006 σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήδη είχε διευκρινίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η έρευνα αποτελούσε τέτοιο κίνητρο και υπήρχαν διάφορα έγγραφα που ανέφεραν την προσέγγιση αυτή. Αν τώρα λοιπόν βγούμε και πούμε ότι η έρευνα δεν αποτελεί κίνητρο, αυτό αποτελεί αλλαγή πολιτική. Αυτό ενδεχομένω να το επιθυμούν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αλλά αυτό θα προαπαιτεί αλλαγή του κειμένου επίπεδου 1. Για το CSA τώρα. Όπως ξέρετε, ούτε οι τεχνικές συστάσει τη ΕΣΜΑ, ούτε τα διάφορα σχέδια τα οποία κυκλοφορούν για τις πράξεις καταξίωση οδότηση, δεν περιλαμβάνουν το τι είναι το CSA. Γιατί δεν είναι η βάση της εργασίας μας αυτής. Η βάση της εργασίας μας είναι να δούμε τι, σε ποιες περιπτώσεις η έρευνα θεωρείται κίνητρο και πότε όχι. Γι' αυτό θέλουμε λοιπόν τη διαφάνεια και το unbundling. Αυτό χρησιμοποιήθηκε στα σχέδια κειμένου. Δεν ξέρω καν τι είναι CSA. Γιατί ορίζεται με διαφορετικό τρόπο στα διάφορα κρατημέλη. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε στην παρούσα φάση το ερώτημα αυτό η βάση των εργασιών μας είναι να ορίσουμε πότε η έρευνα δεν θεωρείται κίνητρο. Για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την απαγόρευση των κινήτρων. Τώρα, σε ό,τι αναφέρεται τα όσα αναφέρθηκαν, σε ό,τι αφορά όσα αναφέρθηκαν για το κόστος. Η τεχνική σύσταση της ΕΣΜΑ ήδη σύστησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τον τομέα αυτό για να είναι ίσοι κανόνες για όλους. Και ασφαλώς ε, θα λάβουμε υπόψη το σχόλιο αυτό σε ό,τι αφορά τα παράγωγα παθονυλών. Βασικό ζήτημα σε ό,τι αφορά τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση αποτελεί το στοιχείο της αναφοράς. Και εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω το εξή. Όταν εξελιγούμε τα ζητήματα αυτά, πολλοί στρέφονται προ το σύστημα των ΙΠΑ. Αλλά είναι διαφορετικέ οι αγορέ μα, είναι οι διαφορετικέ οι διατάξει μα για τις προμήθειες. 28 συμβάσεις ε, στη ΣΥΠΑ όπως αναφέρθηκε, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε χιλιάδες τέτοιες συμβάσεις. Θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη όταν ε, ε, υπολογίζουμε τις διατάξεις και τις απαιτήσει που θα πρέπει να επιβληθούν. Για το σύστημα Tech Internalizer. Τέθηκε το θέμα και το ερώτημα κατά πόσο είναι διμερείς αυτές οι διατάξεις. Το κείμενο σε επίπεδο 1 θεωρεί ότι είναι διμερείς. Και άρα θα πρέπει να τηρήσουμε όσα προβλέπονται στο κείμενο επίπεδο 1. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα του Προέδρου για την ε, εμπορία υψηλής συχνότητας και τον αντίκτυπο στο εθνικό χρέος. Αυτό συζητιέται στο επίπεδο ΕΣΜΑ τη στιγμή που προετοιμαζόταν ε, η τεχνική, τεχνική γνωμοδότηση. Και τότε καταλήξαμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι δεν έπρεπε να δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερο σύστημα για τέτοια ε, για τέτοιες περιπτώσεις εμπορίας υψηλής συχνότητας. Γιατί αυτό πηγάζει άμεσα από το κείμενο επίπεδου 1. Άρα, η ο υπολογισμό από πλευρά τη ΕΣΜΑ θεωρώ ότι λαμβάνει ήδη υπόψη τι διάφορε αγορέ. Και για να κλείσω και συγγνώμη που μακρηγόρησα, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα τα σχόλιά σα, Θα θέλαμε να ακούσουμε και περαιτέρω σχόλια από τα μέλη του Κοινοβουλίου. Ο στόχο είναι να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει συνέπεια μεταξύ επίπεδου 1 και 2 και ότι το επίπεδο 2 θα προβλέπει σαφήνεια νομική και ασφάλεια νομική. Και να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο οι κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα ο κύριος Μέιερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τα μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ να απαντήσω για διάφορα ζητήματα και να δώσω και το λόγο μετά στο Ροντρίγκο για να απαντήσει σε κάποια πιο συγκεκριμένα ζητήματα. Τώρα, για κάποια πιο γενικά θέματα. Ακούσαμε ότι δεν επαρκεί η διαφάνεια που έχουμε και ότι θα πρέπει να υπάρχει προθυμία για πιο οριστικές και σαφείς θέσεις. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο διαφανείς γίνεται. Θα θέλαμε να συνεχίσουμε. Τις συζητήσεις όπως η σημερινή. Έχουμε κάνει τέτοιες συζητήσεις και στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε, αλλά να έχουμε υπόψη ότι είμαστε ένα συμβούλιο 28 μελών. Πολλά από τα ζητήματα τα οποία συζητούμε λοιπόν σήμερα εδώ πέρα είναι ακόμη συζήτηση. Μπορούμε να σας παρουσιάσουμε το τι είναι σημαντικό για τη λήψη αποφάσεων και τι εξετάζουμε, αλλά δεν μπορώ να πάρω οποιαδήποτε οριστική θέση γιατί πολύ απλά αυτό υπόκειται στην έγκριση του Συμβουλίου για το ευρύτερο θέμα των τεχνικών προτύπων για να απαντήσω και στα σχόλια του Μάρκου Φέρμπερ όντω. Σκοπός μας είναι και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει και το τεχνικό φόρουμ τεχνικών προτύπων. Υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής α, εκ των υστέρων. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να πάμε σε αλλαγή πλήρης του επίπεδου 1. Αυτό είναι το πλεονέκτημα το να υπάρχουν τεχνικά πρότυπα. Ανάλογα με τις ε, εξελίξεις στην αγορά μπορούμε να κάνουμε προσαρμογές. Αυτό κατά μέσο όρο παίρνει ένα έτος. Θα ήθελα να υποστηρίξω επίσης το εξή. ότι δεν πρόκειται για πειραματισμό, αλλά όντως χρησιμοποιούμε τα τεχνικά πρότυπα αυτά για να προσαρμοζόμαστε στις εξελίξεις της αγοράς και Αυτό θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή του MIFID. Να κοιτάξουμε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια πριν και μετά την εμπορία. Τονίζουμε ότι αυτό συνάδει με την Ένωση Κεφαλαίου Αγοράς και η ιδέα της διαφάνειας ε, σκοπό έχει να βελτιώσει την ε, λειτουργία της αγοράς ομολόγως, γιατί είναι πολύ διαφορετικές ε, στην φύση τους. Άρα, η τελική πρόταση, όποια και αν είναι, ο αριθμός των ομολογών θα είναι σχετικά μικρός. Μιλάμε για 2.000-2.500 από 15.000 ε, σχετικά αξιόγραφα. Άρα μιλάμε για ένα τμήμα μόνο της αγοράς ομολόγων και για την συμπερίληψή τους στο καθεστώς διαφάνειας. Όπως έχουμε δει στο παρελθόν, έχουμε διαβουλευτεί για το Κόφια και τον Ινδία στην τελευταία έκδοση, στην ε, έκδοση του Δεκεμβρίου. Χρησιμοποίησαμε το κόφια, αλλά όντω να διευκρινίσω ότι εξετάζουμε και τις ε, δύο αυτές ε, εκδοχές της κόφια και της ίδια. Είναι πολύ διχασμένη η αγορά. Είναι πολλοί αυτοί που ένθερμα υποστηρίζουν το κόφια, άλλοι παράγοντες της αγοράς είναι σαφώς υπέρ του συστήματος Ήμπια, άρα θα πρέπει να λάβουμε κάποια απόφαση θα είναι δύσκολο. Δεν μπορώ να σας δώσω οποιαδήποτε οριστική απάντηση, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται ε, ακόμα με έντομο τρόπο. Εν συντομία για την ε, ε, συνοχή μεταξύ MIFID και TRIPS και αντί συγγνώμη, θα πρέπει να πληρούνται οι διατάξεις του MIFID 2, αλλά ξέρουμε ότι οι διατάξεις του USIT δεν είναι α, ίδιες με τις διατάξεις του MIFID σε ό,τι αφορά τις, ε, τα βασικά στοιχεία. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν ε, συντονισμός, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εργαστούμε πιο πολύ στο USIT για τις, ε, τα κίνητρα και την έρευνα. Να συμφωνήσω με αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2010, ε, έρευνα κίνητρο. Αυτό ήταν η γραμμή μας ως έσμα. Και επίσης ε, μείναμε εκτός συζήτηση για τα CSA, γιατί δεν είναι ένας νομικά ορισμένος όρος το CSA. Δεν θεωρήσαμε λοιπόν ότι μπορούσαμε να αποφανθούμε, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ήταν ε, σύμβατα με τις συστάσεις μας στα CSA, αλλά επειδή δεν υπήρχε σωστός ορισμός, δεν μπορέσαμε να αποφανθούμε. Ωρα Βρήκο. Ευχαριστώ. Θα αντιμετωπίσω το θέμα για τα παράγωγα των βασικών προϊόντων. Υπήρξαν πολλά σχόλια από τους περισσότερους βουλευτές οι οποίοι έλαβαν το λόγο για τη γενική ε, ιδέα του 25% είναι 15 εκατοστίες μονάδες. Έχουμε αφιερώσει μεγάλη προσπάθεια στο να βελτιώσουμε το σύστημα αυτό και να το ξανασυζητήσουμε. Δεν έχουμε όμως ε, εντοπίσει ένα καλύτερο σύστημα το οποίο συνδυάζει την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο εύρος των ε, ορίων θέσης, όπως εσείς έχετε καταλάβει και τον πολυμορφό χαρακτήρα των παραγόγων βασικών προϊόντων που αντιμετωπίζουμε και την ανάγκη να υπάρξει εναρμόνιση των καθεστώτων στην Ευρώπη. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν στην προσπάθεια να βελτιώσουμε το σύστημα και είναι σαφές ότι για μερικά συμβόλαια τα οποία δεν έχουν επαρκή ρευστότητα, ακόμα και το 40% της συνολικής αγοράς μπορεί να έχει ένα περιορισμένο όγκο. Κάποιες στιγμές έχετε μακρινές ημερομηνίες τελικής ε, πληρωμής και η κάθε πλευρά έχει ουσιαστικά το 50% της αγοράς. Αν γίνεται αντιστάθμισμα βέβαια δεν θα είναι με στο όριο, αλλά αν όχι θα υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο θα επηρεάσει τις αγορές. Αυτό το οποίο προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε είναι να καθορίσουμε τα κριτήρια που θα πρέπει να εφαρμόσουν οι εθνικές αρμόδιες αρχές όταν βρίσκουν ποιο επίπεδο θα πρέπει να εφαρμόσετε σε κάθε περίπτωση. Είναι γεγονός ότι ορισμένε περιπτώσεις αυτοί οι οποίοι κρίνουν τα όρια κρίνουν επί τη βάση των πιο ε, ακραίες περιπτώσεις όπως παραδείγματος χάρη σε αγορά σπότ για τροφιμικά βασικά προϊόντα με το όριο αυτό του 25%. Εθνικές αρχές λοιπόν θα πρέπει να έχουν μια αρκετά προσεκτική εφαρμογή των ορίων με τρόπο ο οποίο να προσαρμόζεται προς τι ανάγκε της αγορά. Είναι απαραίτητο να κατανοούμε ότι τα όρια αυτά δεν χρειάζεται να είναι στατικά, μπορούν να προ να προσαρμόζονται και να κατεβαίνουν καθώς πλησιάζει η ημερομηνία εκτέλεση του συμβολέου. Πρέπει όμως να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα ότι πολλά από αυτά τα συμβόλαια είναι πολύ χαμηλού ύψους, είναι πάρα πολύ λίγοι συμμετέχοντες, δεν έχουν την απαραίτητη ρευστότητα, γι' αυτό οι εθνικές αρχές χρειάζονται την απαραίτητη ευκαμψία. Υπήρξε και μια συζήτηση, ένα ερώτημα μάλλον από τον κύριο Γίγκολτ, για το, κάσο, για το πόσο ο ορισμός του ίδιου συμβολέου ή όχι <clears throat> θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετικά καθεστώτα και παρεθνικοποιηση για το <clears throat> της αγοράς. Νομίζω ότι εδώ η αντιμετώπιση της ΕΣΜΑ είναι πολύ σωστή. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ακόμα και χωρίς μια νομική ε, εντολή η δράση της ΕΣΜΑ έχει καταφέρει να εξασφαλίσει μεγαλύτερη σύγκληση μεταξύ των ε, εθνικών καθεστώτων ε, το κάνουμε αυτό για τις εξαιρέσεις πριν από το εμπόριο και έχουμε ε, μέχρι στιγμής επιτύχει οι εθνικοί ρυθμιστές να ακολουθούν τις γνωμοδοτήσεις της ΕΣΜΑ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, προς το παρόν συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά μαζί τους για να αποφύγουμε αυτή την επανεθνικοποίηση και την ανάδυση διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. Κάποια περαιτέρω στοιχεία τα οποία αναφέρθηκαν προηγουμένως για τις ε, παράπλευρες δραστηριότητες. Υπήρξε το ερώτημα του κύριου Φέρμπερ ποιος θα καταμετρά τον όγκο της αγοράς, ποιος θα είναι ο παρονομαστής για τα όρια στις, ε, στις συμπληρωματικές ή παράπλευρες ε, διαδικασίες. Φυσικά υπάρχει το πρόβλημα των στατιστικών για το σύνολο της αγοράς, αλλά εμείς προσπαθούμε να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν τους υπολογισμούς αυτούς. Για τις δέσμες ε, συναλλαγών, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα και έχετε διατυπώσει όλες τις ε, σωστές ερωτήσεις για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι για να είμαι πραγματικά ε, ειλικρινής υπάρχει και ένα νομικό θέμα για τις ε, δέσμες ε, συναλλαγών. Το πώς καθορίζεται αυτό, πώς μπορεί να συναρμοστεί αυτό με το επίπεδο 1. Αυτό είναι ένα θέμα που είναι ακόμα εκρεμές σε νομικό επίπεδο. Δεν μπορώ να σας πω πώς θα το κάνουμε, το εξετάσουμε πολύ προσεκτικά, αλλά υπάρχουν κάποιοι νομικοί περιορισμοί σε σχέση με την αντιμετώπιση των ε, δεσμών συναλλαγών, παρά το γεγονό ότι καταλαβαίνουμε ότι είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε το ακατάλληλο καθεστώ και ένα ακόμα θέμα το οποίο δεν συζητήθηκε για τα θέματα των διαφανείων, της αν η προ και μετά τη συναλλαγή τα, η αξιολόγηση διαφάνεια θα πρέπει να έχει το ίδιο κατόφλι. Σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να έχουμε λοιπόν διαφορετικά κατόφλια για, την, ε, ε για τον έλεγχο διαφάνεια πριν και μετά από μια συναλλαγή. Ακόμα προσπαθούμε να βρούμε μια λύση η οποία θα λειτουργεί και η οποία θα βελτιώσει το συνολικό καθεστώ. σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ο πρόεδρος. Ο εισηγητή θα θέλει να κάνει κάποια σχόλια για τη συνέχεια που πρέπει να δώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια μικρά σχόλια όχι επί του περιεχομένου, αλλά επί της διαδικασίας περισσότερο. Καταρχήν, ό,τι και να κάνετε, θα πρέπει να περάσετε από ένα σημείο συμφόρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. <clears throat> Για να αντιμετωπίσετε λοιπόν με σωστό τρόπο αυτό το θέμα, θα γίνει μια συνάντηση απόψε της ομάδος ε, διαπραγματεύσεις του Κοινοβουλίου, εμού και των σχεδόν εισηγητών και θα προσπαθήσουμε να διατυπώσουμε μια κοινή προσέγγιση η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη από την ΕΣΜΑ και από την Κομισιόν για να μπορέσετε να αποκομίσετε την έγκριση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Γιατί αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι έχετε εσείς τη δική σας άποψη και εμείς τη δική μας, εσείς θεωρείτε ότι εσείς έχετε δίκιο και εμείς όχι. Δεν είναι έτσι που δουλεύουν τα πράγματα. Το 2010 ήταν η μύφη η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς εγκρίνουμε την νομοθεσία και όχι εσείς λάβετε υπόψη ότι δεν είναι ένα παιχνίδι που απλώς γίνονται ανταλλαγές απόψεων και ο καθένας κάνει μετά ό,τι, ό,τι θέλει. Πρέπει να συνεργαστείτε και η συνεργασία απαιτεί κοινέ απόψεις. Θα πρέπει λοιπόν να ακούσετε την κοινή άποψη που θα δημιουργήσουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσείς θα πρέπει να ελέγξετε κατά πόσον τελικά οι εφαρμοστικές πράξεις, οι πράξεις κατά εξισιοδότηση, οι κανόνες, οι οδηγίες κατά εξισιοδότηση συναρμόζονται με αυτά τα οποία λέει το Κοινοβούλιο και αυτό περιλαμβάνει και τα δεσμευτικά πρότυπα. Πάρτε το στα σοβαρά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ λέει και ο Πρόεδρος. Η κατεξουσιοδότηση πράξης είναι μια εξουσιοδότηση προς την Κομισιόν να τροποποιήσει μια νομοθετική πράξη στα μη ουσιώδη στοιχεία της και αυτό φυσικά μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, δεν θα μια αυτόματη, θα ήταν μια αυτόματη διαδικασία. Όλοι ξέρουμε λοιπόν τι είναι το ουσιαστικό στοιχείο της νομοθεσίας και το τι δεν είναι και μια κατεξουσιοδότηση πράξη δεν μπορεί να ανατρέψει τα ουσιώδη στοιχεία ενός νομοθετήματος. Ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτές οι τροποποιήσεις αυτών των στοιχείων και αυτό θα πρέπει να υπόκειται σε μια δημοκρατική διαδικασία. Αυτή είναι η κανόνες μας. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία όσο γίνεται και θα ξεκινήσει αυτό με τη συνάντηση των σκιωδών εισηγητών το βράδυ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την τόσο καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων. We move to point 8 of the agenda. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 8 της ημερησίας διατάξεως. So we can Πρόεδρος, να προχωρήσουμε λοιπόν. start. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Ελβικιανίκε, πρόεδρο του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανση, καθώς επίσης ε, και τον Αντιπρόεδρο Λοτινιέμι. Καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας. Είναι η πρώτη δημόσια ακρόαση την οποία οργανώνουμε μετά την τοποθέτησή σας στη θέση του ε, Προέδρου μετά από απόφαση του ε, Διοικητικού Συμβουλίου της 14ης Αυγούστου. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν ε, ευελπιστούμε ότι θα ξεκινήσουμε μία καρποφόρα και επικοδομητική συνεργασία. Να σας πω ότι χτες ε, ε, επετεύχθη η πολιτική συμφωνία όσον αφορά τη συμφωνία η οποία προβλέπεται από το άρθρο 45 του Συμβουλίου Υγείας, συμφωνία με το Κοινοβούλιο, έλεγα. Επομένως ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε σε αυτήν την καλή συνεργασία και θα ξεκινήσουμε και θα συνεχίσουμε μια καλή θεσμική ε, συζήτηση ε, μεταξύ μας. η πρόεδρος ε, κυρία Κιόνιγκ εκλήθη έτσι ώστε να ασχοληθεί με συγκεκριμένα θέματα. Πρώτα απ' όλα ε, ε, ζητήματα εξυγίασης, ας πούμε όπως η περίπτωση της ΕΤΑ. Επίσης, να μας πει που έχουν φτάσει οι συζητήσεις στα πλαίσια του άρθρου 40, 74 ε, συγγνώμη, του κανονισμού. Επίσης, ε, με, ποιους, με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί ο κανονισμός 806, κυρίως όσον αφορά ε, το transfer και mutualization των πόρων. Τέλος, το θέμα του απόρριτου χαρακτήρα ε, των πληροφοριών. Αυτά είναι κάποια θέματα τα οποία εμείς θα θέλαμε να θίξετε, αλλά βεβαίως ε, ε, μπορείτε, κυρία Πρόεδρε, να αναφερθήσετε σε οτιδήποτε σχετίζεται με το Συμβούλιο Εξυγίασης και, το, και τα θέματα τα οποία θεωρείτε ότι καλό είναι να συζητηθούν εδώ. Παρακαλώ πολύ, κυρία Κένικ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έντιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι που είμαι εδώ ενώπιον σας. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από την αρχική μου ακρόαση για να γίνω πρόεδρος της, ε, του, Συμβουλίου, του, του Συμβουλίου του ενιαίου Συμβουλίου Επίλυσης. Τα έξι μέλη μας έχουν ε, αναλάβει τα καθήκοντά τους το Μάρτιο του 2015. Είδα έκτοτε ότι υπήρξε πάρα πολλή εργασία από όλους μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το συμβούλιο αυτό, το ενιαίο συμβούλιο επίλυσης και εξυγίανσης των τραπεζικών φορέων. Μετά από την πρόσκλησή σας, λοιπόν, θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία, όπως φαντάζεστε και εσείς, για να σας δώσω και μία ε, εικόνα της κατάστασης ό,τι αφορά τη δια, την δημιουργία αυτού του Συμβουλίου και στη συνέχεια, όπως αναφέρατε, θα αναφερθώ σε περιπτώσεις ε, επιλύσεως και εξυγίανσης, τα διδάγματα τα οποία έχουμε αντλήσει από αυτά, τα θέματα της εμπιστευτικότητας στη διαδικασία εξυγίανσης και επίσης το Ταμείο Ενιαίας Εξυγίανσης που είναι ένα θέμα στο οποίο θα με βοηθήσει και ο αντιπρόεδρος μας γιατί είναι το δικό του ακριβώς θέμα. Έρχομαι λοιπόν στην ουσία κατευθείαν. Πρώτα απ' όλα μερικές πρακτικές πτυχές. Έχουμε τώρα 60 μέλη του προσωπικού και αυτό περιλαμβάνει 8 μέλη από, το, από την ε, Task Force της Κομισιόν που εξακολουθούν να μας βοηθούν στη δημιουργία του φορέα μας. Έχουμε ιδιαίτερα εξειδικευμένο προσωπικό και μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να έχουμε μια ισορροπία σε σχέση με τα δύο φύλλα και επίσης ισορροπία σε ό,τι αφορά την εθνική εκπροσώπηση. Όπως έχω πει όμως και στο παρελθόν, μπορεί κανείς να προσλάβει μονάχα μέλη του προσωπικού χάρη σε μια ε, ισορροπία στις αιτήσει που γίνονται δεκτές. Αλλά για αυτό το λόγο ζητώ από τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν ότι όταν ζητούμε, κάνουμε μια πρόσκληση για αιτήσει, θα υπάρξει και περισσότερο ενδιαφέρον στα κράτη-μέλη. Οι διοικητικές δομές λοιπόν έχουν δημιουργηθεί και φυσικά εμείς θα πρέπει να στεγάσουμε κάπου το προσωπικό μας και έχουμε βρει ένα ε, μόνιμο κατάλημα στις Βρυξέλλες. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε στις αρχές του 2016 να εγκατασταθούμε εκεί. Η μεγάλη πρόκληση για μας είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε μέχρι το τότε τον Ιανουάριο του 2016 χωρίς να κοιμούμαστε κάτω από γέφυρες τρένων. Προσπαθούμε να βρούμε λοιπόν προσωρινές λύσεις, όπως οποιαδήποτε εταιρεία η οποία ξεκινά από το μηδέν. Εμείς πρέπει να εργαστούμε για τα θέματα αυτά, αλλά συγχρόνως αντιμετωπίζουμε και τα θέματα που πρέπει να, να φέρουμε σε πέραστα. Θα πρέπει να έχουμε ενιαίους κανόνες, ενιαίες διαδικασίες για την εξυγίανση και την διάλυση των πιστοτικών ιδρυμάτων που είναι μέσα στον τομέα αρμοδιότητός μας. Θέλουμε να έχουμε λειτουργικούς κανόνες επί τη βάση και των κανόνων του ESM, του Ταμείου Σταθερότητα σε ό,τι αφορά την διαδικασία εξήγηση και επίλυση τραπεζών. Προσπαθούμε επίση να εντοπίσουμε και να άρουμε τα εμπόδια στο να γίνει το τραπεζικό σύστημα της Ευρώπης πιο εύρωστο και ανθεκτικό. Και φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη και το διεθνές περιβάλλον. Για να μπορέσουμε να επιτύχουμε λοιπόν όλους αυτούς τους στόχους έχουμε δημιουργήσει με απόφαση της ε, Ολομέλειας των Επιτροπών του Ενιαίου ε, Φορέα Επίλυσης, Επιτροπές για την σχεδίαση της εξήγησης και επίλυσης, για την διαχείριση κρίσεων και ένα εγχειρίδιο επίσης για να αντιμετωπίσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες και επίσης για τις ε, συνεισφορές των τραπεζών στο Ταμείο που είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Οι επιτροπές αυτές λοιπόν έχουν ξεκινήσει το έργο τους και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να έχουμε μια σωστή συνεργασία με τις Εθνικές Αρχές εξήγηση και Επίλυσης. Ο στόχος μας είναι να έχουμε το εγχειρίδιο του φορέα μας μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό είναι απαραίτητο και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε πολύ νωρίτερα και για το Ταμείο Εξήγησης και επίλυση θα έρθω αργότερα. Ένα άλλο σημαντικός στόχος για του επόμενου μήνες είναι το έργο μα που συνεχίζεται για τα μνημόνια κατανόηση με διάφορους εμπλεκομένους και ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και επίσης η Συμφωνία συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και φυσικά έχουμε συγγνώμη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα έρθω μετά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη συνέχεια. Ελπίζουμε να έχουμε μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που θα είναι έτοιμη το φθινόπωρο. Η προηγούμενη εμπειρία μας δείχνει ότι αυτό χρειάζεται αρκετές διαπραγματεύσεις. Είναι σαφές ότι ο διαμοιρασμός πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για σκοπούς ρύθμισης είναι πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα και είμαστε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον εποπτικό της μηχανισμό για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και πριν να έχουμε ακόμα τον τελικό κανονισμό για τα θέματα αυτά. Μας το επιτρέπει η νομοθεσία, είναι κάτι το ασφαλές και δεν είναι κάτι που θα σας εκπλήξει όταν σας πω ότι χρειαζόμαστε πληροφορία ήδη στη φάση σχεδίασης της εξυγίανσης και της επίλυσης και όχι μόνο στη φάση που αναλαμβάνουμε επίσημα τις εξουσίες μας για να επιλύσουμε προβληματικά ιδρύματα. Για να είμαι πλήρης, όπως είπε και ο πρόεδρος σας προηγουμένως, η συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ε, Συμβουλίου ε, Ενίας Εξυγίανσης έχουν προχωρήσει πολύ θετικά αυτές οι διαπραγματεύσεις και ελπίζω ότι το ταχύτερο δυνατό θα μπορέσει να υπογραφεί η συμφωνία και από τις δύο πλευρές. Είναι πιο πολύ πρόβλημα επιμελητίας παρά πρόβλημα περιεχομένου αυτή τη στιγμή. Σε σχέση με τη διεθνή συνεργασία, για να έρθω στο θέμα αυτό, συνεχίζονται οι προσπάθειες για να έχουμε ένα μνημόνιο και κατανόησης και με κράτη τα οποία δεν συμμετέχουν και με τρίτες χώρες και κυρίως τις Ηνωμένε Πολιτείες. Και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στα ερωτήματα τα οποία έχετε θέσει εσείς. Έχετε αναφερθεί σε περιπτώσεις εξηγίας και επίλυσης στο παρελθόν. Εγώ θυμάμαι ότι την 1η Μαρτίου που ήταν μία Κυριακή, εμένα πήρα ένα τηλεφώνημα από τους Αυστριακούς συναδέλφους που είπαν ότι ξεκίνησαν ένα μορατόριουμ για το πιστοτικό αυτό ίδρυμα και ξέρετε ότι οι περιπτώσεις αυτές για το 2015 εξακολουθούν να είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα των ρυθμιστών των κρατών μελών βάσει των ε, εθνικών μέτρων εφαρμογής το, το, τραπεζικό, το Τραπεζικό Συμβούλιο είναι ακόμα σε μεταβατικό στάδιο μέχρι το 2016. Κάνουμε το σχεδιασμό για την εξυγένση και επίλυση, αλλά μόνο από το 2016 θα αναλάβουμε πλήρω τα, τα καθήκοντά μας. Στην περίπτωση τη ΧΕΤΑ υπάρχει μια πρόσθετη μνήμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η ΧΕΤΑ δεν έχει άδεια τραπεζικών δραστηριοτήτων και επομένω δεν εμπίπτει στην ε, αρμοδιότητα την, ε, του ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και Επίλυσης. Συγγνώμη. Η ΧΕΤΑ λοιπόν δεν είναι στην αρμοδιότητά μας προς το παρόν για το 2015, ούτε και στο μέλλον θα εμπλέκεται στην αρμοδιότητά μας. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε σε επαφή με τους αυστριακούς συναδέλφους μας και θα εξετάσουμε την περίπτωση αυτή μαζί τους, αλλά όλα αυτά παραμένουν μόνο μέσα στα πλαίσια της άντλησης διδαγμάτων από προηγούμενες περιπτώσεις, τι πρέπει να συμπεράνουμε και τι πορίσματα να αντλήσουμε και πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε για το μέλλον για οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και ιδίως αυτές οι οποίες δεν πέρασαν τα stress test της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με μεγάλη ευτυχία, εμείς είμαστε σε επαφή με τις Εθνικές Αρχές Εξυγένσης και Επίλυσης, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τα σχέδια τα οποία αφορούν τους φορείς αυτούς έχουν δημιουργηθεί. Θα έχουμε φυσικά ένα κατάλογο προτεραιοτήτων για τα θέματα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι οι τράπεζες έχουν σχέδια ανάκαμψης και εξυγένσης και φυσικά το ελέγχει μαζί μας. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εμείς λοιπόν θα πρέπει να συνεργαστούμε γιατί το να υπάρχουν σχέδια, σχέδια εξυγένσης είναι απαραίτητο και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να ευθυγραμμίσουμε τις προτεραιότητές μας ώστε να λειτουργούμε επί τη βάση του ίδιου καταλόγου προτεραιοτήτων. Αυτά ήθελα να σας πω και είμαι έτοιμη να θέσω ε, για το θέμα αυτό να απαντήσω σε ερωτήματα. Έρχομαι τώρα στο θέμα του Ταμείου Εξυγένσης και Επίλυσης. Τους τελευταίους μήνες το Συμβούλιο Εξυγένσης έχει αντιμετωπίσει τις διάφορες ε, δυνατότητες προχρηματοδότησης αυτού του Ταμείου και από ιδιωτικούς και από, από ιδιωτικές και δημόσιες πηγές. Εμάς μας ενδιαφέρει λοιπόν να καλύψουμε αυτή την περίοδο 8 ετών μέχρι την πλήρη χρηματοδότηση του Ταμείου. Επί τη βάση λοιπόν μιας προκατακτικής ανάλυσης που έκανε η ομάδα μας, καταλήξαμε στο ότι, ότι υπάρχουν ιδιωτικές πηγές εξωτερικής χρηματοδότησης καταρχήν, αλλά είναι περιορισμένες σε ό,τι αφορά το μέγεθος και τη διαθεσιμότητά τους. Οι συζητήσει με τους συμμετέχοντες στην αγορά έχουν δείξει ότι <clears throat> οι, οι πιστώσεις που μπορούν να δοθούν από τράπεζες και άλλου άλλους φορείς που είναι υπορρύθμιση δεν είναι ελκυστικές πηγές χρηματοδότησης για πολλούς λόγους. Θεωρούμε λοιπόν ότι λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ μπορεί να προκύψει από τέτοιες πηγές. Η πρόσβαση στην κεφαλαία αγορά, όχι δηλαδή δανειοδότηση από τράπεζε, αλλά πρόσβαση στην κεφαλαία αγορά, υπολογίζεται ότι μπορεί να μας δώσει μεταξύ 5 και 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε αιτήσια βάση, ίσως και μέχρι 25 δισεκατομμύρια και αυτό εξαρτάται από τις ε, οικονομικές συνθήκες και τους νομικούς περιορισμούς η πρόσβαση λοιπόν στην κεφαλαία αγορά θα είναι κάτι το οποίο θα αποτελεί μια πρόκληση λόγω της ε, αδύρυτης πολυπλοκότητος της κατακαιρματισμένης λειτουργίας του Ταμείου μας επειδή δεν υπάρχει επαρκής γνώση σε σχέση με τη λειτουργία του μηχανισμού μας στην αγορά παρά το γεγονός ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το το κάνουμε γνωστό το πώς λειτουργούμε και επειδή βρισκόμαστε ακόμα στη φάση εκκίνησης του, ε, του Ταμείου θα χρειαστεί να δοθεί μια πιστοληπτική αξιολόγηση στο Ταμείο μας και θα υπάρξει και ανάγκη να πιστοποιηθεί ο μηχανισμός συλλογής κονδυλίων. Θα πρέπει να φτέσουμε λοιπόν πολλά ερωτηματικά πίσω από τη διαδικασία αυτή και πιστεύουμε ότι τα πράγματα αυτά θα είναι ρευστά μέχρι το 2016, ίσως το δεύτερο τμήμα του 2016 θα φέρει μεγαλύτερη σαφήνεια. Για να κλείσω λοιπόν, αν <clears throat> πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για δανειοδότηση από το, από το Συμβούλιο, αυτά θα πρέπει να γίνουν στην ολομέλεια του βάση του κανονισμού. Πάμε τώρα στις δημόσιες πηγές χρηματοδότησης. Παρά τις δηλώσεις του Σεπτεμβρίου 20 του ΕΚΟΦΗΝ, βάσει των οποίων θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να υπάρξει γεφυρωτική χρηματοδότηση όταν είναι ήδη δημιουργημένο το Ταμείο μας. Προς το παρόν δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Τους τελευταίους μήνες το Ταμείο Εξυγίανσης και Επέλυσης μαζί με τους διάφορους ευρωπαϊκούς φορείς έχουν εξετάσει τις δυνατότητες για τέτοιες προσωρινές ρυθμίσεις. Εμείς ως ε, ε, Συμβούλιο Επίλυσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση από γραμμές πίστοσης που δίνονται από τα κράτη-μέλη, γιατί με τον τρόπο αυτό θα έχουμε ένα περιθώριο ρευστότητος για το Ταμείο Επίλυσης και Εξυγίανσης, θα βοηθήσουν να ανυψώσουν το προφίλ τους στις κεφαλαιαγορές και θα εξασφαλίσουν την διαθεσιμότητα των κονδυλίων όπου και όταν χρειάζονται. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το έργο για την πρακτική εφαρμογή αυτής της λύσης μετά από την απόφαση που ελήφθη σε πολιτικό επίπεδο, ώστε να έχουμε αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, να έχουμε δημόσια χρηματοδότηση από την 1η Ιανουαρίου του 2016. Και ας πηδήξω προς το ερώτημα της συγκεκριμένης, της συγκεκριμένης εφαρμογής του, του κανονισμού 806 κάθετος 2014. Βάσει των πληροφοριών μας. Είναι κάπως λυπηρή η ιστορία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μόνο δύο κράτη-μέλη έχουν κυρώσει την διακυβερνητική συμφωνία και κάποια άλλα προβλέπουν να το κάνουν στο άμεσο μέλλον. Και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανοικοδόμησης, μόνο 7 κράτη-μέλη έχουν την ERD. Μόνο 7 κράτη-μέλη έχουν ε, εγκρίνει και εφαρμόσει την ERD. Και θα ήθελα λοιπόν να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία να ζητήσω τη δική σας υποστήριξη για να υπενθυμίσετε στα κράτη-μέλη που το έχουν λησμονήσει και δεν έχουν εφαρμόσει αυτή τη συμφωνία την, ε, το νομοθέτημα αυτό ότι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσει την ε, λειτουργία του φορέα μας. Είναι η εργαλειοθήκη μας αυτό το νομοθέτημα. Δεν θα μπορούμε να έχουμε έναν αρμονισμένο μηχανισμό που να λειτουργεί εάν δεν μα δώσει τα κατάλληλα εργαλεία. Τελευταίο λοιπόν σχόλιο που θέλω να κάνω το θέμα της εμπιστευτικότητας. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί είτε πρόκειται για κάτι που έχει να κάνει <clears throat> με την ε, εποπτεία ή την εξυγίανση. Είναι μεγάλη σημασία η διαδικασία αυτή και γι' αυτό η ταξινόμηση και η ανταλλαγή δεδομένων είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του φορέα μας και των εθνικών εμπλεκομένων. Για να εξασφαλιστεί λοιπόν αυτή η εμπιστευτικότητα αυτό πρέπει να γίνει με το μνημόνιο κατανόηση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να αναφέρεται και στις συμφωνίες μη αποκάλυψης που θα συνάπτονται με τους εμπλεκόμενους φορείς σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμεί θα αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό στην επικείμενη συμφωνία συνεργασία που δεν έχει ακόμα διατυπωθεί, αλλά είναι υποσυζήτηση με την Κομισιόν και νομίζω ότι έχουμε μια κοινή κατανόηση και από τι δύο πλευρέ για το θέμα αυτό, για την ανάγκη να υπάρξει επιμερισμό ε, μυστευτικών πληροφοριών και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν ήδη κάποιε διατυπώσει στην διαθεσμική δεν ξέρω αν είναι διαθεσμική, αλλά εν πάση περιπτώσει τη συμφωνία αυτή μεταξύ ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ε, Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης. Ελπίζω λοιπόν θα μπορέσουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα μαζί μέσα στα πλαίσια του πλαισίου εμπιστευτικότητας που καλύπτεται από το κανονισμό μας και πιστεύω ότι αυτός είναι ένας πολύ καλός κανονισμός όταν πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς για θέματα εμπιστευτικότητος και γι' αυτό νιώθω μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα μπορέσει να καλυφθεί το θέμα αυτό. Ε, νομίζω ότι έχω καλύψει όλα τα θέματα και τώρα είμαι έτοιμη να απαντήσω οποιοδήποτε ερώτημα που ίσως έχετε είτε εγώ είτε ο Τίμ για το Ταμείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ εκτενή παρουσίαση και για το γεγονός ότι απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα που έχουμε θέσει για τα συγκεκριμένα ζητήματα που μας απασχολούν και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι όλοι μας θα πρέπει να πιέσουμε στα εκάστοτε κράτη-μέλη για την πλήρη εφαρμογή του BRD και φυσικά και του των διατάξεων του Ταμείου Εξυγίανσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να εφαρμοστούν. Θα δώσω το λόγο στον πρωτομιλητή. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κ. Μπάλτσα, αγαπητή κυρία Κόνιγκ, χαίρομαι ιδιαίτερως ε, που μπορώ να ακούσω σήμερα τα σχόλιά σας ε, ως ε, πρόεδρο της υπηρεσίας εξυγίανσης. Δεν είναι σίγουρα εύκολο να δημιουργηθεί από το τίποτα ένα τέτοιο οργανισμό όπω το Σύμβουλο Εξυγίανση. Έχετε πάρα πολλά να κάνετε. Πρωτού ε, η υπηρεσία σα μπορεί να αναλάβει τα καθήκοντά σα το επόμενο έτο. Αλλά είμαι βεβαίω ότι βρίσκεστε σε καλό δρόμο. Τρει ερωτήσει έχω να κάνω. Καταρχά, μιλήσατε για τι ε, νέε δομέ που πρέπει να δημιουργηθούν για τη νέα υπηρεσία αυτή. Θα ήθελα να μα πείτε, αυτέ οι δομέ πώς θα διαμορφωθούν με λίγο μεγαλύτερη ακρίβεια και τους επόμενους ε, μήνες κατά την οικοδόμηση της υπηρεσίας σας. Τι θεωρείτε ότι θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη πρόκληση. Ποιες θα είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες δηλαδή. Δεύτερη ερώτηση για τη μεραβική σας εργασία. Θα είναι σημαντική η ανταλλαγή δεδομένων και η συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Πώς λοιπόν πιστεύετε ότι θα δημοκρατεί αυτή η εθνική συνεργασία και κοιτώντα τις εθνικές αρχές εξυγίανσης και τους εθνικούς επόπτες, μπορώ να περάσω και στην τρίτη ερώτησή μου κατευθείαν. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για τους πρώτους μήνες της συνεργασίας σας, πώς διαμορφώθηκαν. Είπατε ότι αναμένετε να γίνουν πολλές, ε, πολύ ενδιαφέροντες γύρια διαπραγμάτευσης με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πώς εκτιμάτε λοιπόν την συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με την ε, Εποπτική Αρχή. Ευχαριστώ πολύ. απάντηση. Να απαντήσω στα γερμανικά. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Καταρχάς, οι δομές. Ποιες είναι οι βασικές δομές και ποια είναι τα βασικά προβλήματα. Είμαστε καινούργια επιχείρηση, ξέρετε. Άρα κάνουμε βλέποντας και κάνοντας σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε. Ο Τιμ θα συμφωνήσει μαζί μου. Και τα πιο βασικά θα πρέπει να τα οργανώσουμε εξ αρχή. Η πρόσληψη του προσωπικού αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση. Ναι, ούτε εμεί έχουμε καλό καφέ, λέει ο κ. Βέρμπερ. Όχι, όχι αυτό που είπα για τα θεμελιώδη και χρειώδη που πρέπει να οργανώσουμε και τον καφέ, το παίρνω πίσω. Βασική λοιπόν πρόκληση είναι το πώς θα φτιάξουμε μια σωστή ομάδα. Προσλαμβάνουμε άτομα με υψηλά κίνητρα, αλλά με πολύ διαφορετικό πολιτισμικό και πολιτιστικό υποβατρό Για να υπάρχει λοιπόν μια ισορροπία στην ομάδα, να μπορούμε όλοι να ε, μιλάμε, αν θέλετε, με τους ίδιους όρους και να εννοούμε το ίδιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μια νέα υπηρεσία. Θα τα πετύχουμε. Και το κτίριο αποτελεί ένα βασικό ζήτημα. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να μετακομίσουμε το 2016. Αλλά αναπτυσσόμαστε ταχύτατα. Και δεν μας φτάνουν τα γραφεία που έχουμε. Άρα αναζητούμε και προσωρινές λύσεις για την διάμεση περίοδο. Και επίσης ένα βασικό θέμα είναι να ξεκινήσουμε για θέματα περιεχομένου σε ό,τι αφορά τα διοικητικά, το διοικητικό ναι. σκέλο. Ε, ήμασταν τυχεροί γιατί είχαμε την Task Force τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί είναι άνθρωποι που ξέρουν τι διαδικασίε στο έπακρο και μπορούν να μα βοηθήσουν να τι εφαρμόσουμε μέσα στον τρόπο. Αυτά είναι τα τεχνικά ζητήματα, τα τεχνικέ προκλήσει. Και επίσης άλλο θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε σχέδια για 150 τράπεζες, ε, πολλές εξ των οποίων είναι και μεγάλες μέχρι τέλη του έτους, άρα θα πρέπει να γίνει κάποια επιλογή, να μπουν προτεραιότητε και σε κάποιο βαθμό, και έτσι θα περάσω στην τρίτη σας ερώτηση, έχουμε θέματα με τις εθνικές αρχές εποπτείας και εξυγίανσης, γιατί όπως ξέρετε η αλλαγή της αρμοδιότητας θα γίνει το 2016. για παράδειγμα για την ελάχιστη ευθύνη οι σχετικές διατάξεις θα τεθούν από το 2016. Αλλά σαφώς οι εθνικές αρχές μας ζητούν να τους ε, αναφέρουμε ποια θα είναι η πολιτική μας για να τη χρησιμοποιήσουν στα σχέδια εξυγίανσης, να ξέρουν προς τα ποια κατεύθυνση θα κινηθούν. Άρα Έχουμε πολλά να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τις χώρες. Έχουμε κάποιε χώρες ε, που έχουν ήδη ξεκινήσει εγκαίρως και έχουν ε, αρχές εξυγίανσης ε, μεγάλου μεγέθους και κάποιες με μεγάλη εμπειρία, αλλά έχουμε και χώρες οι οποίες τώρα συστήνουν τις υπηρεσίες αυτές. Αυτό με τη σειρά του τι σημαίνει. Ότι αντίθετα με τον ενιαίο εμποπτικό μηχανισμό δεν έχουμε την ε, πολυτέλεια να πούμε ότι αν δεν συμφωνήσουμε κάτι για φέτος, θα πούμε ότι θα το κάνουμε όπως το κάναμε πέρσι, όπως το έκαναν δηλαδή οι εθνικές αρχές ε, το περασμένο έτος, γιατί δεν υπάρχει τέτοια θέση. Η συνεργασία λοιπόν με τις εθνικές αρχές έως τώρα λειτουργεί καλά. Νομίζω ότι υποβοηθάτε και από τις επιτροπές που συστήσαμε και τη συνεργασία μας μαζί της δεν είναι δηλαδή ότι το ε, ενιαίο Συμβούλιο εξυγίανση ξέρει τα πάντα. Ιδιαίτερα εδώ στις Βρυξέλλες. Μία επιτροπή που επικεντρώνεται στη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών και ημών. Έχει ήδη καταθέσει την ιδέα να ακολουθήσουμε το ίδιο μοντέλο όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δηλαδή, να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τη συνεργασία με το ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης και με, τα εθνικά, με τις εθνικές αρχές. Τέλος, και με την ε, ΕΚΤ. Με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Η συνεργασία είναι εξαιρετική, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ποιο είναι το διακύβευμα αλλά παράλληλα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι μια με πολύ μεγάλη οργάνωση και όλα παίρνουν χρόνο. Για παράδειγμα, για το πολύ απλό ζήτημα της ανταλλαγής πληροφοριών και πολύ απλά κάποιες φορές δεν έχουμε και χρόνο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Για να δώσουμε το λόγο σε όλους τους ομιλητές θα πρέπει να τηρήσουμε τα τέσσερα λεπτά για κάθε έρωτα απάντηση. Άρα σας παρακαλώ συνάδελφοι, ένα-ενάμιση λεπτό μάξιμου η ερώτησή σας για να έχουμε τρία λεπτά για την απάντηση. Η Ελίδα Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά μια ναι, και εσείς ε, επίσης επιλέξατε να μας μιλήσετε αγγλικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε και σας και την ομάδα σας για την εργασία που έχετε κάνει. Μας απασχολεί πάρα πολύ, ε, με τα, μας απασχολούν πάρα πολύ τα στοιχεία τα οποία μας δώσατε όσον αφορά το ε, επίπεδο μεταφοράς του PRT. Ε, είναι ανησυχητικό που το BRD, το οποίο θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί και ενσωματωθεί μέχρι το Δεκέμβρη του 2014, ε, έχει τελικά ενσωματωθεί μονάρα στην νομοθεσία 7 κρατών μελών. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Λυπούμαστε επίσης γιατί ε, και μονάχα δύο κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει σε, στην ενσωμάτωση άλλων διαδικασιών πολλά σας περιμένουν από τις αρχές του επόμενου χρόνου και επομένως ερωτώ ποια είναι η επαφή σας με την Κομισιόν και το Συμβούλιο και φυσικά και το Κοινοβούλιο, ε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να ε, ασκήσετε πολιτική πίεση γιατί δεν είναι πάρα πολύ ε, χρόνος, έχουμε φτάσει ήδη στα μέσα του τρέχοντος έτους και επομένως ε, θα πρέπει να γίνει ε, μία κατά κάποιο τρόπο εντελεχής μελέτη της κατάστασης έτσι ώστε ε, να δείτε ακριβώς με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να προχωρήσετε. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη όσον αφορά τα backslope που πάντα ήταν προβληματικό. Δεν ε, ήταν πολύ σαφής η άποψή σας και θα ήθελα να μου εξηγήσετε πρώτον ποιο, που, έχει φτάσει η συζήτηση ε, για τις δυνατότητες του ESM που είχε ξεκινήσει ε, σαν ε, βοήθημα ας πούμε της δυνατότητας που έχει ο μηχανισμός εξυγίανσης και τι γίνεται σε σχέση με τις μεμονωμένες πιστοτικές γραμμές από τα κράτη-μέλη είναι ένα πάρα πολύ περίπλεκο ε, ε, ζήτημα και αν επιλέξετε τις, αυτές τις γραμμές θα είναι ακόμα πιο περίπλοκο. Στην πρώτη σας ερώτηση ε, απαντάω θετικά, συμφωνώ. Χρησιμοποιούμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε έτσι ώστε να πούμε ότι η BRD θα πρέπει οπωσδήποτε να ενσωματωθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα στις χώρες μέλη. Τώρα, Εκτός από το να κάνουμε έκκληση σε όλους, δεν έχουμε άλλα μέσα συγκεκριμένα. Αλλά για να είμαστε και ε, δικαιοί, η Κομισιόν ε, πραγματικά έχει ενστερνιστεί την προσπάθεια και έχει ήδη ε, ε, κοινοποιήσει σχετικές επιστολές στις χώρες οι οποίες δεν έχουν φτάσει στην τελική φάση και επομένως και η Κομισιόν χρησιμοποιεί τη δική της εργαλειοθήκη για να προωθήσει. Ε, νομίζω ότι παρότι πήρε πολύ χρόνο μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Ε, δεύτερον, εμείς ως SRB όταν ξεκινήσαμε μας ζητήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με τις ε, διάφορες ε, εναλλακτικέ. Και εμείς καταλήξαμε ότι οι, ε, οι, ιδιωτικές λύσεις ναι είναι περιορισμένου εύρους όντως αλλά ε, είδαμε και διάφορες εναλλακτικέ όσον αφορά την δημόσια τις δημόσιες λύσεις, λύσεις με το δημόσιο τομέα ε, και ε, φτάσαμε σε κάποιες για την ώρα ε, και για τα επόμενα 8 χρόνια καταλήξαμε σε κάποιες λύσεις κατακαιρματισμένες, κατατμημένες στον δημόσιο όμως τομέα. Ωστόσο θα το ξαναδούμε το, το ζήτημα αυτό και αναφερθήκατε βεβαίως στον ESM. Από από τον τρόπο με τον οποίο κατανοώ εγώ την κατάσταση, ο ESM δεν μπορεί άμεσα, απευθείας να δανείσει τα SRM, αλλά, αλλά ε, νομίζω ότι τα ίδια τα κράτη-μέλη, το Συμβούλιο θα πρέπει ε, να πάρει την τελική απόφαση. Εμείς έχουμε ε, υποβάλει κάποια πρόταση και περιμένουμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κυρία, Καν, ε, και κυρία που ήρθατε ενώπιον μας σήμερα. Το ερώτημά μου έχει να κάνει με τον στόχο της ε, μείωσης του κόστους για τον ε, φορολογούμενο σε σχέση με όλες αυτές τις δραστηριότητες του ελέγχου και της επίλυσης. Αλλά έχετε μια σειρά από εξαιρέσεις σε σχέση με την, ε, από την εφαρμογή του bail Και επίσης έχει, υπάρχει μια εξαίρεση για τις ε, υποχρεώσεις, για τις υποχρεώσεις έναντι φορέων που έχουν διάρκεια λιγότερο από 7 μέρες. Γιατί λοιπόν γίνεται αυτή η προνομιακή μεταχείριση στο άρθρο 140 για ορισμένους φορείς και για τις ε, υποχρεώσεις έναντι κάποιων φορέων. Υπάρχει μια συγκεκριμένη εξ, ε, εγγύηση για, όλες, για όλους αυτούς τους φορείς και αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο κόστος που πρέπει να υπομειστεί ο φορολογούμενος για την εξυγίανση και την επίλυση μιας τράπεζας. Μήπως οι περιπτώσεις αυτές που έχουν να κάνουν με την χρονική διάρκεια των 7 ημερών θεωρείται μια κρατική εγγύηση για διατραπεζικές ε, συναλλαγές. Μια έμεση λοιπόν ε, εγγύηση η οποία δεν οδηγεί σε κάποιο κόστος για τις ε, τράπεζες αυτές. Αυτό δεν πρέπει να μείνει κάτι το οποίο θα είναι αδιαφανές για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Και επίσης αυτό το είδος εγγύησης, έμεσης εγγύησης δίδει ε, ουσιαστικά στις τράπεζες κίνητρα να προβούν σε περισσότερες συναλλαγές ή μπορείτε αλλιώς να το εξαιρέσετε αυτό, να το να το αποκλείσετε. Βάσει του άρθρου 140 και, το, και σε ό,τι αφορά το bail-in. Για μένα αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στο άρθρο 140 που λέει ότι εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι γίνεται αυτή η διαδικασία του bail-in και ότι θα πρέπει να προηγηθεί οποιοδήποτε άλλου μέτρου το οποίο θα λυθεί. Το ενιαίο Ταμείο Επίλυσης μαζί με τα κατημέλη συνεργάζεται για να μπορέσει να εξασφαλίσει ότι θα μπορεί να είναι πραγματικά λειτουργικό το bail-in σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα εδώ είναι το θέμα ότι υπάρχει μια κατηγορία πιστωτών οι οποίοι έχουν ε, κάποια προηγούμενα δικαιώματα, κάποια προτεραιότητα ικανοποίηση δικαιώματο, όχι μόνο αυτό που αναφέρεται στις 7 μέρες αλλά και οι καταθέτες και δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία ε, διάκριση μεταξύ των, ε, ε, αυτο, των πιστωτών. Το πιο σημαντικό εδώ είναι στην περίπτωση επίλυσης να υπάρξει και κάποια σκέψη για το ποιος είναι ο βαθμός στον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι πιστωτές που έχουν χαμηλότερη προτεραιότητα και πώς μπορούν να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Εγώ νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό. Παραμένουν ακόμα ανοιχτά ερωτήματα. Το ερώτημά σα σε σχέση με την ε, προνομιακή θέση των ε, ετοιμάτων που είναι διάρκειες, έχουν χρονική διάρκεια λιγότερο από 7 ημέρες. Αυτό δεν είναι, ε, είναι κάτι που αφορά τη διατραπεζική αγορά. Εμείς δεν βλέπουμε κάποια τροποποίηση με αυτά τα οποία ισχύουν. Εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτό θα μπορούσε να απαντηθεί βάσει των στοιχείων που έχουμε. Ίσως η Κεντρική Τράπεζα να έχει καλύτερα στοιχεία για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Στόιρερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Κιόνιγκ και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ε, δηλώσεις σας, για την παρουσίαση σας εδώ να σας ευχαριστήσω και εσάς και την ομάδα σας. Έχω τις εξής συγκεκριμένες ερωτήσεις. Καταρχάς, πείτε μας, αντιμετωπίζετε προβλήματα και συγκεκριμένα όρια σε ό,τι αφορά την απόκτηση ειδικού προσωπικού ή βρίσκεται στους κατάλληλους εμπειρογνώμονες. Δεύτερη ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τις έντονες ε, οξύες κρίσεις που παρουσιάζονται σε κάποιες χώρες. Ανακύπτει το ερώτημα ότι ενδεχομένως να υπάρξουν στο εγγύς μέλλον υποθέσεις ε, στην ε, Ευρώπη που θα υπερ θα επέβαλαν υπερβολικό άχθος ε, στο Συμβούλιο σας. Πώς λοιπόν θα μπορούσατε να ανταποκριθείτε στις απαιτήσει αυτές. Και επιτρέψτε μου και την ερώτηση την εξή. Πώς ε, αξιολογείτε τις εξελίσεις ε, με την κατάσταση στην Ελλάδα στο πλαίσιο αυτό. Μάλιστα, και τώρα θα μιλήσω πάλι στα αγγλικά, λέει η κυρία Κιόνιγκ, για την πρόσληψη. Προς το παρόν νομίζω ότι δεν έχουμε έλλειψη υποψηφίων με τα κατάλληλα προσόντα. Πρέπει να πω ότι έχουμε και μια καλή εκπροσώπηση στα βιογραφικά από τον αντιτικτικό τομέα, όχι μόνο από το δημόσιο τομέα. Είναι, υπάρχουν προκλήσεις ε, στα θέματα ισότητας φύλων, ίσης εκπροσώπησης εθνικότητων, όταν έχουμε πιο, πολλές, ε, ε, πιο πολλά βιογραφικά ανδρών, είναι δύσκολο να κάνουμε επιλογές για να υπάρχει ισότητα άνδρων και γυναικών ή ίση προσώπηση χωρών. Άρα ενθαρρύνω την αποστολή βιογραφικών. Ο κίνδυνος ε, να πνιγούμε, να πλημμυριστούμε από καθήκοντα όταν ξεκινήσουμε τον Γενάριο του 2016. Ελπίζω πως όχι. Όλοι μας, οι επόπτες, ε, όλοι έχουμε εργαστεί σκληρά για να πάνε όλα καλά. Αλλά αν κάτι πάει στραβά το δεύτερο ήμιση του έτους, θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Σε εμά επαφείεται και στους υπόπτες, προκειμένου να υπάρξει μια καλή αρχή. Αυτό που είναι πιο σημαντικό, και εδώ δράτω με τις ευτερίες να πω το εξής, δεν φαίνεται λογικό όλοι να έχουν δικαίωμα να εξηγένονται από εμάς. Όταν μια τραπέζα έχει προβλήματα, καταρχάς η τράπεζα πρέπει να το επιλύσει. Αν όχι, περνάει σε διαδικασία πτώχευσης. Αυτό είναι το επόμενο λογικό βήμα. Και μόνο αν η εξυγίανση θα καταλήξει σε καλύτερο αποτέλεσμα για το κοινό και για όλους, θεωρείται ότι αποτελεί μία πιθανότητα, μία δυνατότητα. Και αυτό, όπως είπε η κυρία Φεραίρα, θα ισχύσει. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να τα περάσουμε αυτά το 2016 για την Ελλάδα. Όλοι παρακολουθούμε τις ειδήσει και πάντα λέω ότι οι ελληνικές τράπεζες ζουν σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Αλλά αυτό που είναι πολλά υποσχόμενο είναι ότι είναι ενεργός, είναι πολύ ενεργή η ομάδα, μικρή η ομάδα εξυγίανσης, δεν είναι μεγάλη, αλλά έχει εμπειρία σε εξυγίανση τραπεζών και είμαστε σε στενές επαφές με τους Έλληνες συναδέλφους. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ο κ. Βιέγκας. Ε, Ευχαριστώ. Έχω τρία ερωτήματα. Διάβασα το έγγραφο που έχει διανεμηθεί και βλέπω ότι αφορά, περί, αφορά μοναχα 55 τράπεζες. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο τα στοιχεία για αυτές τις 55 τράπεζες είναι αντιπροσωπευτικά της γενικής κατάστασης. Ή έχουμε απλώς μια έρευνα που αφορά τις τράπεζες που βρίσκονται στις καλύτερες καταστάσεις. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν κατά πόσο είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα του γενικού συστήματος αυτό το δείγμα των 55 τραπεζών που την χάνουν άμεσης εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο ερώτημα αφορά το βαθμολόγιο αυτό που προσπαθεί με αντικειμενικά στοιχεία να καταμετρήσει τον κίνδυνο αφαιρεγκιότητος για τις ε, τράπεζες και την ανάγκη παρέμβασης του μηχανισμού επίλυσης. Δεν ξέρω, θα ήθελα να ξέρω πώς θα γίνεται αυτό. Θα υπάρχει μια περιοδική έκθεση, μια περιοδική αξιολόγηση για κάθε μία από τις τράπεζες και αν αυτά τα στοιχεία θα δίδονται στη δημοσιότητα θα είναι στη θέση του, διάθεση του Κοινοβουλίου και τρίτο για το Μπέιλιν και τις εξηγήσεις που έχετε αναφέρει. Και ένα από αυτά είναι το κατά πόσο η κατάρρευση μιας τράπεζας μπορεί να είναι συστημικός κίνδυνος. Μα θα ήθελα εδώ να ξέρω τι γίνεται για να γίνεται μια αντικειμενική αξιολόγηση του κινδύνου επιμόλυνσης ή του κινδύνου συστημικότητος ενός ιδρύματος για να εξαιρεθεί από τη διαδικασία Μπέιλιν. Ευχαριστώ. Νίσο, με το πρώτο ερώτημα. Τα 75 δις ε, είναι η αξιολόγησή μας βασιζόμενη στο 1% εγκυημένων καταθέσεων και ε, θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι με τις προσπάθειες που κάνουμε τώρα ότι θα υπάρξει ομοιόμορφος μηχανισμός ε, ε συμβολής δεν ε, βλέπω να υπάρχει ε, οποιαδήποτε εύνοια από τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Ο μηχανισμός ε, εξυγίανσης ε, και ε, η εκ των προτέρων αξιολόγηση με αυτό είναι κυρίως ο στόχος των προγραμμάτων εξυγίανσης που έχουμε, τα οποία τουλάχιστον εν μέρει απαντούν και την τελευταία σας ερώτηση, είναι εστιασμένα στην διασυνδεσιμότητα των τραπεζών, στο ίχνος που έχει η κάθε τράπεζα και οπωσδήποτε στην φερεγγιότητα εν τέλει της τράπεζας σε σχέση με την σημασία τους. Δηλαδή ε, ε, δεν θα είναι το ίδιο, η ίδια ε, η αντιμετώπιση μιας μικρής τοπικής τράπεζας με μια μεγάλη διεθνική διασυνδεδεμένη τράπεζα τώρα τα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ε, είναι οπωσδήποτε ε, ε, θέματα τα οποία σχετίζονται με εξυγίανση <coughs> διασυνοριακή και διεθνική. Εκεί βεβαίως θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους άλλους ομολόγους μας των άλλων των διαφόρων χωρών. Αλλά μία ε, συγκεκριμένη πτώχευση οπωσδήποτε μπαίνει σε, σε λογική ε, γενικότερη. Ο Σβέν ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω γερμανικά κυρία Κόνικ. Χαιρόμαστε που βρίσκεστε και πάλι μαζί μας. Ωστόσο, δύο ερωτήσει έχω να σας κάνω. Καταρχάς θα ήθελα να μου πείτε τα μεγάλα οι μεγάλες ε, τράπεζες που επηρεάζουν το σύστημα, όπως αναφέρατε. Για αυτές θα υπάρχουν σαφείς κατευθύνσεις για το τι περιμένετε από αυτές προκειμένου να, είναι, να έχουν την ε, δυνατότητα να εξηγιαθούν. Θα δώσετε καθοδήγηση. Έχει νόημα, για παράδειγμα, να είναι ε, να υπάρχει δυνατότητα εξυγίανση μια τράπεζα που θα περιλαμβάνει πάνω από χίλιε εντότητε. Θα πρέπει να υπάρξει πρώτα μια αναδιάρθρωση τη τράπεζα αυτή. Δεύτερη ερώτηση. Για μια α, συνέντευξη που κάνατε στο Handelsblatt που με εξέπληξε και παραθέτω στην ερώτηση, κυρία Κόνιγκ, όλε τι ημέρε, όλες τα θέματα αυτά όλες τις, ε, σήμερα όλοι μιλάνε για την Ελλάδα και για την πτώχευσή της. Ε, αυτή την ερώτηση απαντάτε, θα πρέπει να τη θέσετε στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά μου φαίνεται ότι έχουν στονέψει τα χρονικά περιθώρια. Χρειαζόμαστε πάρα πολύ οσιοδεξία για να πιστέψουμε ότι εγκαίρω θα μπορεί να βρεθεί μια λύση. Και εκ των υστέρων μιλάτε για το ELA, για τον ε, αρρωγή ρευστότητας και σε ό,τι αφορά τι ελληνικέ τράπεζε. Αναρωτιέμαι κατά πόσον είναι υπεύθυνο να κάνετε τέτοιες δηλώσεις, τέτοιες, εποχές, τέτοιες εποχές, τέτοιες στιγμές. Κατά πόσον αυτό συγκαταλέγεται και στην εντολή σας. Η συζήτηση που γίνεται για το απόρριτο των ε, εγγράφων του Κοινοβουλίου και όπου υπάρχει αμφιβολία για το κατά πόσον υπάρχει εμπιστευτικότητα στην αντιμετώπιση των ε, ε, εγγράφων στο Κοινοβουλίο. Μήπως θα έπρεπε να το θέσουμε αυτό το θέμα και για σας ε, τέτοιες ε, στιγμές μου. Προκαλεί έκπληξη λοιπόν αυτή η συνέντευξη και θα ήθελα ε, να ξέρω κατά πόσον όντως δώσατε τις δηλώσεις αυτές, γιατί δεν πιστεύω τα μάτια μου σχεδόν. Η απάντηση. Να... Να απαντήσω στην πρώτη σας ερώτηση για τις ε, μεγάλες που επηρεάζουν συστημικά Σίγουρα θα υπάρχει καθοδήγηση για το τι μπορούν να κάνουν. Αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουν και μαθήματα για το σπίτι, αν θέλετε. Μια φορά καθήκονται. Στη συζήτηση για το TILAC, για παράδειγμα, θα επικεντρωθούμε και σε θέματα συστήματων IT, fit for person, ε, διαφάνειας, διαφορετικά ζητήματα στα οποία και αναφερθήκατε δεν έχει να κάνει αυτό με ποιο τύπο τράπεζα ενδείχνεται, αλλά με το ποιες λειτουργίες είναι κρίσιμες και μπορούν εύκολα να απονομωθούν σε έναν όμιλο, αν μπορεί να υπάρξει διάκριση του ομίλου. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Ναι, ναι, λοιπόν, θα υπάρξει καθοδήγηση, δημόσια συζήτηση τώρα. Κάποια θέματα είναι γνωστά, νομίζω. Για την ε, συνέντευξη στο Handelsblatt, στη Handelsblatt. Η συνέντευξη, αν την εξετάσατε σε βάθος, ήταν για τα καθήκοντα της SRB. Ήταν μια γενική ερώτηση αυτή. Ναι, όπως συνήθως η απάντηση ήταν πιο εκτενής. Αλλά όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε από το πρίσμα της συζήτησης. Ο κ. Γκίγκολτ, πιστεύετε ότι είναι υπεύθυνο να κάνετε τέτοιε δηλώσει και πώ σχετίζεται με την εντολή σα. Αυτό το ερώτημα έθεσα. Η απάντηση. Νομίζω ότι το νόημα τη συνέντευξη ήταν για το SRB. Η απάντηση αυτή ήταν μια απάντηση γενική ε, φύσεως, ότι θα πρέπει κανείς ε, να είναι αισιόδοξο για να πιστεύει ότι θα βρεθεί λύση. Ήταν μια γενική παρατηρήση την οποία δικαιούται ο καθένα να κάνει, θεωρώ. Σα ευχαριστώ. Δεν έχω δει το κείμενο τη ε, συνέντευξη. Ε, θα σα παρακαλέσω μετά να μα το στείλετε και θα μπορέσουμε να το ξανασυζητήσουμε στην ομάδα εργασία για την Τραπεζική Ένωση. Μάρκο Βάλι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε Ανίκα που ήρθατε σε αυτήν την προκαταρτική εκφάση να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Εγώ έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την επιλογή του προσωπικού. Με ποιο τρόπο κινείστε. Ε, κάνετε περισσότερες μόνιμες συμβάσεις ε, ή ε, συγκεκριμένου χρόνου έχετε ε, επιλέξει προσωπικό το οποίο θα δουλέψει για πολύ καιρό μαζί σας. Επίσης, ε, ε, όσον αφορά το προσωπικό που προτείνουν οι χώρες είναι με endorsement ή ε, με πιο ποιοτικά ας πούμε κριτήρια. Ε, επίσης σε περίπτωση ας πούμε κολοσσών τραπεζικών Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank κτλ. Πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε την περίπτωσή τους. Πρόκειται για τράπεζες οποίες τα τελευταία χρόνια ε, προτίμησαν τις κερδοσκοπικές ε, ε, κινήσεις και επιχειρήσεις στην αγορά και όχι μονάχα και όχι κυρίως την παραδοσιακή τραπεζική πίστη. Να πούμε ότι η Deutsche Bank απέτυχε στα τελευταία stress test της Άνοιξης και να υπενθυμίσουμε ότι εδώ πρόκειται για έναν οργανισμό που διακατέχει 55 ε, δις ε, μόνο σε παράγωγο. Ευχαριστώ. Απάντηση. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα ε, να απαντήσω το θέμα για το προσωπικό. Ναι, τώρα εμείς προτείνουμε, προσφέρουμε ε, συμβόλαια περιορισμένου χρόνου, ωστόσο το προσωπικό αυτό αργότερα μπορεί να γίνει μόνιμο. Ε, από τα 60 άτομα, 8 ε, προέρχονται από την Task Force της Κομισιόν, αλλά 8 ε, είναι εθνικοί εμπειρογνώμονες που μας έχουν σταλεί και ευχαριστούμε τα κρατη που τους έστειλαν για να μας, τους, για να μας βοηθήσουν ε, και οι υπόλοιποι είναι προσωπικό το οποίο έχουμε προσλάβει ε, εμείς. Πάντα θα έχουμε κάποιους εθνικούς εμπειρογνώμονες, αλλά βασιζόμαστε κυρίως πλέον ε, στο δικό μας προσωπικό. Ε, στην ερώτησή σας μπορεί το σύστημα να ανταποκριθεί ε, και να διασφαλίσει ότι ακόμα και μεγάλες κολυσίες τράπεζες μπορούν να εξηγιανθούν Νομίζω ότι θα απαντήσω ε, με μετριοπάθεια λέγοντας παρόλα αυτά ότι τουλάχιστον πολύ καλύτερα από το παρελθόν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ε, τέτοιου είδους ε, θέματα. Βεβαίως, εάν ένας από τους μεγάλους βιομηχανικούς κολοσσούς αντιμετωπίζει προβλήματα, πάλι θα το καταλάβουμε. Το ίδιο ισχύει και για τις τράπεζες. Το θέμα είναι να γίνουν πιο φερέγγιες οι τράπεζες, να γίνει πιο διαφανές το ε, σύστημα, κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκαναν ε, και οι συνάδελφοι των, ε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκεφτόμαστε λοιπόν ότι θα είμαστε σε καλύτερη θέση και κατά αυτή την έννοια βλέπω πάντα με αισιοδοξία την κατάσταση. Ευχαριστώ. Η Μπάρμπαρα Κάπελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Κιόνικ για την παρουσία σας και για αυτά που είπατε βέβαια η Ελλάδα είναι ένα επίκαιρο θέμα και φυσικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μας δήλωσε χθε ότι η, κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρήσει τις ελληνικές τράπεζες σε επίπεδο φερεγγιότητος και λειτουργικότητος. Εσείς έχετε μιλήσει για μια δυνατότητα επίλυσης και εξήγευσης των ελληνικών τραπεζών. Αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο, κάποια συμφωνία για τα θέματα αυτά. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του κεφαλαίου των τραπεζών αυτών προέρχεται από συνεισφορές φορολογουμένων. Και επομένως νομίζω ότι αυτά που είπατε δεν εφαρμόζονται. Δεν μπορεί λοιπόν είπατε, βάσει αυτών που είπατε, δεν θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνεχίσει να δίνει ρευστότητα στις τράπεζες αυτές. Υπάρχει το πρόβλημα της τράπεζας HETA στην Αυστρία που υφίσταται αυτόρα μια διαδικασία εξυγίανσης και ήδη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία από την 1η Μαρτίου 2015 για να σταματήσουν οι πληρωμές και να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ε, επίλυσης της τράπεζας αυτής μέχρι το Μάιο του 2016 βρέθηκε να υπάρχει ένα κενό κεφαλαίων, ένα χάσμα 4 μέχρι 7,6 δισεκατομμυρίων στο, στον ισολογισμό της τράπεζας αυτής, η οποία συνδέεται με προηγούμενες τράπεζες όπως η Υποάντρια που είχαν εμπλακεί σε κερδοσκοπικές δραστηριότητες ελέγχθη από το Υπουργείο Οικονομικών της Αυστρίας ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω βοήθεια προς την τράπεζα αυτή και θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσης της τράπεζας αυτής βάσει του αυστριακού δικαίου και θα πρέπει να καταθέσει τον ισολογισμό της ώστε να γίνει η, η απαραίτητη διαδικασία ελέγχου που δεν προδιαγράφεται να είναι ιδιαίτερα θετική. Τίθεται εδώ το θέμα λοιπόν της ε, αστικής ευθύνης και του bail-in σε σχέση με το μηχανισμό του bail-in. Αναφέρεται ότι θα πρέπει να εξαιρεθούν από την ε, ε, εγγύηση μεγάλη καταθέτηση. Το ερώτημά μου είναι, σε σχέση με τα θέματα της ευθύνης, πώς θα κάνετε την λειτουργία του bail-in λειτουργική και δεύτερον, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία με πιο γρήγορο τρόπο για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα, λέει η κυρία Κένιγκ, να σας πω ότι δεν είπα στην ε, συνέντευξή μου ότι πρέπει να υπάρξει εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών. Είπα ότι αν υπάρξει πρόβλημα και αυτό ισχύει για όλες τις ε, χώρες και για την Ελλάδα, στην Ελλάδα οι τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα αναλάβουμε την ευθύνη για αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2016. Για το θέμα της ΧΕΤΑ στην Αυστρία δεν είμαστε ούτε τώρα ούτε θα είμαστε και από του χρόνου αρμόδιοι για το θέμα αυτό. Είναι στα χέρια των εθνικών αρχών. Εμείς είμαστε σε επαφή με τις αυστριακές αρχές και μέσα στα πλαίσια της ε, αντιμετώπισης της διαδικασίας της ΧΕΝΤΑ και της Άντρια, της υποάντρια, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει μονάχα είναι τα διδάγματα τα οποία μπορούμε να κλείσουμε από την ιστορία αυτή και όταν πρόκειται για το άρθρο 44, μία από τις κύριες, ένα από τα κύρια εγχειρήματα που πρέπει να, αναλάβουμε είναι το εγχειρίδιο για την ε, αφαιρεγγιότητα και εκεί θα πρέπει να εξασφαλί... θέλουμε να εξασφαλίσουμε ποια είναι τα κατώτερα όρια για τις ε, επιλέξιμες ε, υποχρεώσεις που θα πρέπει να συμμετάσχουν στο bail Ο στόχος μας είναι να υπάρχει ίση μεταχείριση όλων των πιστωτών και θέλουμε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε λειτουργικά να εξασφαλίσουμε αυτόν τον στόχο και φυσικά να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια ιεραρχία πιστωτών μεταξύ των πιστωτών. Και τώρα ξαναγυρίζω στα και ξαναγύρισα στα γερμανικά χωρίς να το καταλάβω. Έχουμε Έχει ολοκληρώσει και ο πρώτο γύρο ε, πολιτικών ομάδων. Θα ήθελα λοιπόν να είμαι πιο αυστηρό. Ε, ένα, ένα μισή λεπτό για την ερώτηση, δυόμιση λεπτά για την απάντηση, γιατί έχουμε ψηφοφορία μετά. Κύριο Ζάλμπα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω για την παρουσία σα την κυρία Κιόνικ αναφερθήκατε στην ε, κατάταξη σε επίπεδο ποιότητας των διαφόρων ευρωπαϊκών τραπεζών. Θα ήθελα να ξέρω αν θεωρείτε ότι έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Επίσης, ποια είναι η σχέση σας με τις αρχές επίλυσης και εξυγίανσης τρίτων χωρών. Ξέρουμε ότι υπήρξε κάποια βελτίωση στις σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά φαίνεται ότι με τη Λατινική Αμερική και τις Ασιατικές χώρες τα πράγματα δεν έχουν προχωρήσει. Και τέλος, Υπάρχουν κάποιες εθνικές αρχές οι οποίες λαμβάνουν ήδη κάποια μέτρα χωρίς να υπάρχει συνεννόηση με τις ευρωπαϊκές αρχές. Είμαστε σε ένα έτος μετάβαση το 2015. Μήπως θεωρείτε ότι οι αρχές επιλύσεως θα πρέπει να στείλουν κάποιες κατευθυντήρες γραμμές στις εθνικές αρχές και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή αυτών των κατευθυντήρων γραμμών. Ευχαριστώ πολύ να σταθώ πρώτα για την ε, μείωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης ορισμένων τραπεζών από την Standard Poor's. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ε, ψηφοφορίας του Κοινοβουλίου που είπε ότι οι πιστοληπτικοί οργανισμοί θα πρέπει να μειώσουν την υποστήριξη για τα κρατικά υπόλογα. Ε, ομόλογα αυτό δείχνει ότι πράγματι πιστεύουν και οι αρχές πιστοληπτικής αξιολόγηση από τον Μπέιλιν. Θεωρώ ότι αυτό είναι θετικό. Εγώ δεν πρόκειται τώρα να κρίνω αν είναι επαρκή η αξιολογήση τους ή όχι. Δεν είναι δικό μου θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα των διαπραγματεύσεων με τις τρίτες χώρες. Έχουν ξεκινήσει αυτές οι διαπραγματεύσεις, προχωρούν βήμα-βήμα. Έχουμε αρχίσει να συνεργαζόμαστε με τους ομολόγους μας στις ΗΠΑ που είναι πολύ σημαντικό θέμα δεν θεωρώ ότι έχουμε αρχίσει πραγματικά συζητήσεις με λατινοαμερικανικές χώρες, αλλά θα γίνει αυτό <clears throat> στο μέλλον. Έχουμε απλώ ένα κατάλογο θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και τώρα για τις κατευθυντήριες γραμμές <clears throat> προσπαθούμε να συνεργαστούμε όσο μπορούμε καλύτερα με τις εθνικές αρχές εξυγένσης και επίλυσης και όπως σας είπα πηγαίνει καλά αυτά και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κατευθυντήριες γραμμές για αυτές αλλά θα πρέπει να κατανοήσετε ότι είναι ο τέταρτο μήνα ύπαρξή μα Δεν μπορούμε να επιτύχουμε λοιπόν να γίνει αυτή η διαδικασία πριν από το καλοκαίρι. Ευχαριστώ. Η Περβάνος Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Που ήσασταν ανάμεσά μας και σα εύχομαι και κουράγιο για την ίδρυση τη υπηρεσία σα όπω μα τα περιγράψατε τα πράγματα. Η υπηρεσία σα, λοιπόν αποτελεί τμήμα ενό πακέτου και λείπει ένα πυλώνα στο πακέτο αυτό, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι τη στιγμή που το Συμβούλιο Εξυγίανσης ξεκίνησε, είχαμε συνείδηση ότι έπρεπε να υπάρξει και ένα τρίτο πυλώνα, αυτό τη εγγύηση των καταθέσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει και επικρατεί μεγάλη ανησυχία, γιατί η ιδέα αυτή τη εποπτεία και τη εξυγίανση πλέον έχει οριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά για να υπάρξει απόφαση που θα επηρέαζε ένα καθώς μέλος συγκεκριμένα μια τράπεζα, η ευθύνη της εγγύησης των καταθέσεων θα παρέμενε εθνική αρμοδιότητα. Είναι μια στρέβλωση αυτή λοιπόν στο νέο αυτό σύστημα που φτιάχνουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα καθήκοντα της είναι δύσκολα και βλέπουμε ότι προτείνονται άλλοι δρόμοι, άλλες ε, μέθοδοι για την εναρμόνιση της ε, εγγύησης των καταθέσεων, αυτό που γίνεται σε ό,τι αφορά την ένωση των κεφαλαγορών. Κάποιοι άλλοι προτείνουν να περάσουμε σε ένα σύστημα όχι εγγύησης καταθέσεων, αλλά ε, ε, διαβεβαίωσης των ε, εγγύησεων. Πώς εκτιμάτε λοιπόν την πρόταση αυτή και σε τι βαθμό πιστεύετε ότι είναι σημαντικό εδώ είμαι, εδώ μπροστά εδώ εδώ, γιατί με ψάχνετε. Σε τι βαθμό λοιπόν πιστεύετε ότι αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά για σας για να είναι μεγαλύτερη η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία της ίδιας σας της υπηρεσίας, του ίδιου του συμβουλίου σας. Είναι σαφές ότι η Τράπεζα και η Τραπεζική Ένωση υποτίθεται ότι θα είχε τρεις πυλώνες. Οι δύο βασικοί πυλώνες λοιπόν υπάρχουν το σχέδιο εγγύησης ε, των καταθέσεων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα αρμονισμένο σύστημα. Αν υπάρχει ένα αρμονισμένο σύστημα σε εθνικό επίπεδο, ακόμα καλύτερα. Κατά πόσο προκαλεί τώρα αρνητικές επιπτώσεις στο ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα στην Τραπεζική Ένωση. Δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι δεν προκαλεί αρνητικέ συνέπειε, αλλά σίγουρα θα πρέπει να προσέξουμε. Thank you. Next. Σας ευχαριστώ πολύ, Μάρκος Φέμπερ. Σας ευχαριστώ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομα. Στην προηγούμενη εβδομάδα η EBA έκανε τεχνικές ε, συστάσεις και δημοσίευσε τη σχετική έκθεση για την δημιουργία του Συμβουλίου Εξηγένσης και προβλέπει ένα περιθώριο για το ελάχιστο όρο στόχο. Θα ήθελα λοιπόν το, κατά πόσο ισχύει το 1% για την αρχή ή για το τέλος της φάσης οργάνωσης και κατά πόσον έχει νόημα να υπάρξει αύξηση του ελάχιστου ορίου αυτού. Δεύτερον, για το πώς ε, ε κατανέμονται οι αρμοδιότητες στο περιθώριο αυτό. Ε, ποια θα είναι η κατανομή, ε, φτάνει το 1% και κατά πόσον έχει νόημα στην αρχή της φάσης προγραμματισμού να υπάρχει μεγαλύτερη συνεισφορά για να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή. Είναι πάρα πολύ έγκυρο το ερώτημα αυτό. Έχουμε αρχίσει ήδη να εργαζόμαστε σε σχέση με την Επιτροπή μας για τις ε, συνεισφορές. Όταν θα έχετε το Ταμείο Επίλυσης και Αξιγίωσης, θέλετε τα χρήματα να μπουν στο Ταμείο το ταχύτερο δυνατό. Απλώς αυτή τη στιγμή ε, αξιολογούμε τις προτάσεις της ε, τραπεζικής, Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής για τα θέματα αυτά και θα ακολουθήσουμε μετά από αυτή την αξιολόγηση. Ήταν πολύ ανοιχτή η απάντηση γιατί δεν έχουμε καταλήξει σε τελική απόφαση σε σχέση με τη χρηματοδότηση αυτή. 8 χρόνια για να μπορέσουμε να φτάσουμε το 100%. Αλλά τότε η αγορά θα έχει καταλάβει ποια είναι η ερμηνεία σας των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, λέει ο κύριος Φέρμπαρ. Θέλουμε μέχρι το φθινόπωρο να λύσουμε το πρόβλημα αυτό, λέει η κυρία Κιόνικ. Ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος λέει το θέμα αυτό τώρα βρίσκεται στα χέρια της Κομισιόν και περιμένουμε από την Κομισιόν να περάσει στο επόμενο επίπεδο και κατά τη διαδικασία αυτή ελπίζουμε ότι θα ζητηθεί και η δική μας γνώμη. Ελπίζουμε ότι η Κομισιόν θα περατώσει το δεύτερο επίπεδο και θα δράσει και θα κάνουμε την εφαρμογή από τη βάση της αποφάσης της Κομισιόν. Μπορούμε να πούμε γενικά ότι το έγγραφο της ΕΜΠΑ, της Τραπεζικής Αρχής, έχει σωστά εντοπίσει την ανάγκη για να υπάρξει το ε, κατώτερο επίπεδο του Ταμείου των 55 δισεκατομμυρίων ευρώ δηλαδή και να γίνει η καλύτερη δυνατή συλλογή των συνεισφορών, να υπάρξει μια σταθερή ροή συνεισφορών ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί η συλλογή αυτών των 55 δισεκατομμύριων ευρώ που είναι η βάση της λειτουργίας του, του Ταμείου. Ο Πέτερ Ζήμαν είναι ο επόμενος Ευχαριστώ κύριε Κιόνιχ έχετε εξηγήσει την δυσαρέσκειά σας γιατί πολλά κρατημέλη δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει και κυρώσει την οδηγία για την ανάκαμψη και την επίλυση. Ας πούμε ότι είναι κάποια που είναι μικρά ή μεγάλα. Ε, τι θα γίνει σε ένα, αν σε ένα από αυτά τα κράτη-μέλη υπάρξει ένα μεγάλο πρόβλημα εξυγίανσης και επίλυσης Παρά το γεγονός λοιπόν ότι αυτά τα κράτη δεν θα έχουν κυρώσει αυτή την ε, ε οδηγία, τι θα γίνει. Θα πρέπει ο φορολογούμενος να παρέμβει και να αναλάβει το βάρος. Επίσης το 2016 θα αναλάβετε την ευθύνη για ένα μεγάλο αριθμό τραπεζών. Πιστεύετε ότι τα κράτη-μέλη αυτά τα οποία δεν θα έχουν, δεν έχουν κυρώσει αυτή την ε, οδηγία θα πρέπει να το κάνουν το ταχύτερο δυνατό και επίσης για τις πληρωμές στο Ταμείο Επίλυσης που βλέπετε τις δυσκολίες για τα 11 αυτά κράτη-μέλη τα οποία πρέπει να συμβάλλουν στο ταμείο αυτό θα υπάρξει κάποια επίπτωση ή δεν θα υπάρξει επίπτωση στην ταχύτητα με την οποία θα καλυφθούν τα χρήματα του ταμείου. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με το πρώτο θετικά νέα είναι ότι όλα τα κράτη, αυτά τα κράτη-μέλη ε, έστειλαν ε, έναν απεσταλμένο ειδικό στην Ολομέλεια, ε, τη δική μας, για να δουλέψει μαζί μας. Δεν ξέρω, έστω, βέβαια το να μην υπάρχει νομική βάση μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα. Ξέρετε και και εσείς ότι η οδηγία ενδεχομένως θα είναι άμεσα εφαρμόσιμη αλλά ίσως είναι και ολυθυρός αυτός ο δρόμος Ωραία. Ε, το θετικό στοιχείο πάντως είναι ότι τα κράτη-μέλη, νομίζω όλα αυτά τα κράτη-μέλη έχουν ξεκινήσει να δημιουργούν την απαραίτητη υποδομή οποτεδήποτε δεν υπήρχε ήδη ε, πληρωμές στο Ταμείο. Θα πρέπει να ξαναδείτε, θα πρέπει οπωσδήποτε η διακυβερνητική συμφωνία να ε, αρχίσει να υλοποιείται. Θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν, να κάνουν δηλαδή την πληρωμή τους ε, στο Ταμείο και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Γκρουμαν Μάρκα. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και για την ε, παρουσίαση. Εδώ είμαι, κυρία Πρόεδρε. Ε, ένα γενικό ερώτημα ποια είναι η άποψή σας ε, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει γενικότερα η εικόνα. Έχουμε γνώση εμείς κάποιων διαφορών, γιατί άλλωστε έχουμε νομοθετήσει για πολλές από αυτές, αλλά θα ήθελα τη δική σας άποψη. Την άποψή σας λοιπόν σχετικά με τον ε, τρόπο με τον οποίο ε, η αφαιρεγγιότητα των τραπεζών έχει ε, μεγαλώσει ή πόσο έχει μικρύνει ο κίνδυνος επιμόλυνσης στο σύστημα. Ακόμα δεν έχει μεταφερθεί η νομοθεσία σε όλες τις χώρες, αλλά όταν θα έχει μεταφερθεί και ενσωματωθεί, πώς νομίζετε ότι θα έχει αλλάξει το τοπίο. Ευχαριστώ πολύ. Απάντηση. Πάντα είναι δύσκολο να δώσει κανείς συγκεκριμένες πληροφορίες. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ε, υλοποίησης των ε, των ε, διαφόρων νομοθετημάτων, λαμβάνοντας υπόψη και την διαφορετική στάση που είχαμε όσον αφορά τις μεγάλες τράπεζες τουλάχιστον στις περισσότερες χώρες ε, να δημιουργήσουν ειδικά ταμεία αντιμετώπισης προβλημάτων, θεωρούμε ότι η αντοχή των τραπεζών και η φερεγγιότητά τους έχει ενδυναμωθεί. Πάντως και το ίδιο το σύστημα είναι πολύ πιο διαφανές και σε καλύτερη κατάσταση, αλλά ακόμα πολλά πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τελευταία ερώτηση, Χώνας Φερνάντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία Κρόνικ. Θα ήθελα να ε, επιμείνω στην ερώτηση που έκανε προηγουμένως ε, η κυρία Μπερέσε σχετικά με το συνδυασμό των ταμείων ε, εγγύσεων και την εγγύηση των καταθέσεων μέσω, αυτού, μέσω του, Ταμείου Εγγυήσεων των καταθέσεων αλλά και αυτού του ενιαίου Ταμείου εξυγίανσης ε, πρόεδρος. Ε, θα έχουμε τρία λεπτά διακοπή για να προετοιμαστούμε για την ε, ε, ψηφοφορία. Επιτρέψτε μας εντωμεταξύ όμως να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας γιατί αλλιώς είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος Φερνάντες. Ε, έλεγα ότι δεν καταλαβαίνω γιατί το Ταμείο ε, Εξυγίανσης ε, δημιουργείται από ένα ποσοστό των καταθέσεων των πιστοτικών ιδρυμάτων, ενώ καλείται να καλύψει στην ουσία το υπόλοιπο του παθητικού των τραπεζών και όχι το, τις καταθέσεις οι οποίες καλύπτονται από τις εθνικές προστασίες. Με κάποιο τρόπο τρόπο δηλαδή οι τράπεζες ε, συμβάλλουν στην προστασία των καταθέσεων, συμβάλλουν και στο Συμβούλιο Εξυγίανσης ε, ε, αλλά τελικά θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο ε, οι, οι, οι τράπεζες εν τέλει συμβάλλουν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Εγγύησης. Πάντως νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε λίγο το σύνολο των εγγύων και των διασφαλίσεων του χρηματοπιστωτικού συστήματος γιατί ξέρουμε ότι αυτά τα ιδρύματα είναι αυτά τα οποία βρίσκονται στο κέντρο του κυκλώνα αυτή αυτής της ε, κρίσης. Ε, ε, δεν σας απασχολεί ότι στην ουσία διαρκώς χρηματοδοτούμε το, το χρέος με τον τρόπο αυτό. Επίσης κάτι άλλο στα πλαίσια των διαβουλεύσεων αναφέρθηκε ότι οι κυρώσεις που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, ε, ε, στα πλαίσια της αρμοδιότητας που έχει ως επιβλέπουσα αρχή μπορεί να εφαρμοστεί και στο Ταμείο Εξυγίασης. Θεωρείτε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εξελιχθεί σωστότερα το Ταμείο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στην πρώτη σας ερώτηση. Η αναφορά των συνεισφορών στο Ταμείο ε, που θα λαμβάνεται από, τα ασφαλισ... από τις ασφαλισμένες καταθέσεις είναι πολιτική νομίζω απόφαση και οπωσδήποτε είναι κάτι ε, το οποίο θα μπορούσε να αντικατασταθεί από κάτι άλλο. Πάντως είναι πιο πολιτική η συζήτηση. Τώρα, ε, υπερφορτώνουμε το σύστημα με τον ε, μηχανισμό εξυγίανσης, ε, με, τον, με το Εθνικό Σύστημα Προστασίας Καταθέσεων, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Καταθέσεων, νομίζω ότι αυτό γίνεται έτσι ώστε να υπάρχει να υπάρχει ασφάλεια των καταθέσεων και αυτό βεβαίως δεν μπορεί να είναι δωρεάν. Δηλαδή πληρώνουμε το κόστος για ένα πιο ασφαλές σύστημα. Ε, δεύτερη ερώτηση, δεν κατάλαβα πολύ καλά την αγγλική μετάφραση. Δηλαδή λέτε ότι οι κυρώσεις ε, τις οποίες ε, θα έχει θα επιβάλλει η Κεντρική Τράπεζα ή οι ρυθμιστικές αρχές θα μπορούσαν ε, να ε, δημιουργήσουν ένα προηγούμενο ή να χρησιμοποιηθούν για το ενιαίο Συμβούλιο Εξυγείας. ενδιαφέρουσα ιδέα, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κιόνι και το Συμβούλιο το ενίο Συμβούλιο εξυγίανση και Επίλυσης για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Θα έχουμε και μια νέα ανταλλαγή απόψεων τον Οκτώβριο. Μέχρι τότε θα έχουμε ψηφίσει τη συμφωνία αυτή μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και πιστεύω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε μια πολύ καρποφόρα ε, θεσμική συνεργασία.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 So, dear colleagues, I think Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες. Όπως ξέρετε, η πρώτη ψηφοφορία είναι η νέα διαβούλευση Κύριε Δεμάζη, ήθελα να θέσω για τα πρακτικά ότι έχω χάσει την ε, κάρτα ψηφοφορίας και θα πρέπει να το κάνουμε Χωρί κάρτα. Ποιοι δεν έχετε κάρτα. Όλοι το ίδιο πρόβλημα έχετε. Ο κ. Σούρτανσου. Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω αναβολή της ψήφου για την έκθεση αυτή. καταρχά γιατί ο κατάλογος ψηφοφορία έφτασε στι 2 το πρωί και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το συζητήσουμε με τους συναδέλφους τα θέματα της ψηφοφορίας και κατά δεύτερον επειδή ζητήσαμε να ψηφιστούν ξεχωριστά 27 ψηφοφορίες λιγότερο από 5 εξετάστηκαν υπάρχουν θέματα που είναι πολιτικώς ευαίσθητα και δεν καλύπτονται τους συμβιβασμούς και νομίζω ότι δεν είναι έτοιμος ο κατάλογος της ψηφοφορίας θέλω λοιπόν να ζητήσω αναβολή της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος να απαντήσω δύο διαφορετικά πράγματα το θέμα της ε, μη κάλυψης των τροπολογιών αυτό είναι μία απόφαση που έλαβα βάσει της, ε, του καταλόγου δεν πρόκειται να αλλάξει σε περίπτωση αναβολής. Καταλαβαίνετε δεν σας αρέσει, αλλά ε, εξαρτάται από το πώς ερμηνεύουμε τις ε, τροπολογίες για την ε, ψηφοφορία. Εγώ προτείνω επίσης σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, ψηφοφορίας πιστεύω ότι θα πρέπει να ψηφιστεί. Αν το θέλετε επισήμω, να το ψηφίσουμε. Αλλά τώρα θα ψηφίσουμε τις πληρωμές. Στο θέμα των πληρωμών για τις πληρωμές. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Για το θέμα της πληρωμής λοιπόν. Στο 9 της ημερήσιας διάταξης. Νέα διαβούλευση με το άρθρο 73 του κανονισμού για τις ε, υπηρεσίες πληρωμών. Ο εισηγητής κύριος Ταγιάννης έχει το λόγο. Ένα λεπτό το πολύ όμως σας δίνω κύριε Ταγιάννη το κόστος ε, ε, του κατακαιρματισμού των, ε, της αγοράς αυτής κοστίζει 1% του ΑΕΠ. Το, το κόστος με, τη, με τις νέες υπηρεσίες πληρωμής οπωσδήποτε θα δημιουργήσει ένα νέο πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τις αγορές αλλά και για τους καταναλωτές. Ε, το Κοινοβούλιο έχει υπεραμεινθεί με, με τεπιτάσεως όλων των επιλογών ε, του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ τον ε, συνάδελφο Φέρμπερ που ήταν πρόεδρος των τριγωνικών διαλόγων. Ευχαριστώ πολύ και όλους τους συναδέλφους, Σάντοους και τα Πάρα πολύ ωραία. Είναι όντως ένα πάρα πολύ σημαντικό νομοθέτημα. Θα ψηφίσουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Να κάνουμε πρώτα μία δοκιμή έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι όλα πάνε καλά. Δοκιμή λοιπόν άρχεται. Okay, the route is closed. Πέρας. Ο κύριος Καράς. Α, δεν έχετε κάρτα. Ποιοι δεν έχουν κάρτα, ο κύριος Δεμάζη, ο κύριος Καράς. Κανείς άλλος. Οι υπόλοιποι είστε στην τάξη και φυσικά η γραμματεία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ε, και τον αριθμό των μελών των πολιτικών ομάδων. Μάλιστα, μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στην ψηφοφορία του συμφωνημένου κειμένου για τις υπηρεσίες πληρωμών στην ιστορική αγορά. Έναρξη ψηφοφορίας παρακαλώ. Μία, δύο ψήφοι παραπάνω από το ΕΛΚ αν υπολογίσουμε και στον κύριο Κάρας. Άλλη μία ψήφος ε, υπεράριθμη από το ΕΛΚ. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Και τώρα έχουμε μισό λεπτό. Τώρα να περάμε στο διαδικασία. Έχουμε την έκθεση Μπερές για ψηφοφορία. Υπάρχει έτοιμα για αναβολή, αν σωστά κατάλαβα. Ε, υποστηρίζουν οι συνάδελφοι αυτό το αίτημα. Μπορούμε να ψηφίσουμε για το αίτημα αναβολής. Μπορώ να ζητήσω να μιλήσει ένας υπέρ, ένας κατά, εφόσον το επιθυμείτε. Ναι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση. Άκουσα τα θέματα που έθεσε ο κ. Ουρτάσουν για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν στη διαδικασία αυτή. Και εμείς έχουμε μια παρόμοια ανησυχία. 15 τροπολογίες έχουν μπει στους συμβιβασμούς, αλλά δεν πιστεύουμε ότι οι τροπολογίες έχουν οποιαδήποτε σχέση με τους συμβιβασμούς που τελικά συμφωνήθηκαν και ότι οι συμβιβασμοί που θα ψηφιστούν ουσιαστικά δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τις τροπολογίες. Άρα, θα ήθελα να υπάρξει αναβολή βάσει του ότι δεν ήταν σωστή η διαδικασία για τις τροπολογίες μας και ε, επειδή αυτές που κατέθεσε και ο κ. Ουρτάνσαν είναι ξεχωριστές και δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τους συμβιβασμούς. Δεν ξέρω βάσει ποιου κανόνα μπορώ να επικαλεστώ την αναβολή. Ούτε ξέρω ποιοι κανόνες σας επιτρέπουν ή δεν σας επιτρέπουν να αποφασίσετε από αυτό. Μάλιστα, είναι σαφές, είναι πάρα πολύ σαφές, λόγια, ο Πρόεδρο, μπορώ να παταδίσω. Αλλά δεν θα γίνει συζήτηση από αυτού, είναι σαφές το αίτημα, έχετε την απάντασή μου η τροπολογία ενδεχομένω να καταπέσει για δύο λόγους. Πρώτος λόγος, γιατί καλύπτεται από ένα συμβιβασμό ή γιατί είναι αντίθετος με το συμβιβασμό. Αλλά αν εγκριθεί λοιπόν το κείμενο του συμβιβασμού, καταπίπτει η τροπολογία. Γι' αυτό λοιπόν δεν ψηφίζονται κάποιες τροπολογίες ή σε κάποιες περιπτώσεις ψηφίζονται. Αυτό είναι θέμα ευκαιρία του εισηγητή. Μπορείτε να το ελέγξετε. Έτσι έχει ο κατάλογο ψηφοφορία λοιπόν. Δεν θα γίνει συζήτηση από αυτό. Έτοιμα αναβολή τη ψήφου. Αν κάποιο συνάδελφο θέλει να υποστηρίξει το αίτημα αυτό, ο κύριο Τόιερ. Ναι, εμεί θα θέλαμε να υπάρξει αναβολή, αλλά για άλλο λόγο. Έχουμε 75 σελίδε για ψηφοφορία, στο κατάλογο ψηφοφορίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσουμε στις 12.30 και έχουμε και συναδέλφου που έχουν να πάνε στη Γενική Γραμματεία. Μα ε, συντομέστε λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος. Δεν έχουμε συζήτηση να κάνουμε συζητήσει. Δεν θα τελειώσουμε στην ώρα μας και θέλουμε βολή. Μάλιστα είναι σαφές λοιπόν το αίτημα. Την άλλη φορά να προβλέψουμε πιο πολύ χρόνο λοιπόν για τόσο μεγάλη ψηφοφορία. Μάλιστα σαφέστατο. Και βεβαίως να είστε όλοι σύντομοι. Όλοι ήταν σύντομοι. Δεν ξέρω ποιο θέλει να μιλήσει κατά τη αναβολή τη ψήφου. Κανεί. Δεν είναι τέτοια παρέμβαση. Να ψηφίσουμε, ο κύριο Λούκε. Έχετε κάτι επιπρόσθετο να πείτε, μην επαναλάβετε τα ίδια. Ναι, με επιτρέψτε μου να πω αυτά που θέλω να πω. Υποστηρίζω το αίτημα των συναδέλφων για την αναβολή τη ψήφου και έχω και έναν επιπρόσθετο λόγο. Γιατί μου φαίνεται ότι. I don't let you finish. The request is... Δεν σα επιτρέπω να ολοκληρώσετε. Το αίτημα είναι για αναβολή της ψηφοφορία. Ο, ο, ο κανονισμός προβλέπει μία παρέμβαση υπέρ, μία κατά. Όλοι μπορούν να φέρουν ένα επιπρόσθετο λόγο. Ακούσαμε δύο επιπρόσθετους λόγους για αναβολή. Τώρα θα ψηφίσουμε για την αναβολή ή μη. Δεν χρειάζεται. Δεν προβλέπεται την διαδικασία. Ο κύριος Μπάρτς. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου ότι πιστεύω ότι θα πρέπει να να σας πω ότι πιστεύω ότι πρέπει να μπορεί να μιλάει κάποιος, να ολοκληρώνει. Το κατά πόσο αυτό αλλάζει κάτι είναι άλλο θέμα. Αλλά δεν μου αρέσει η διαδικασία αυτή. Συνάδελφοι από διαφορετικές ομάδες να θέλουν να παρουσιάσουν τους λόγους που τους αφορούν και να μην τους αφήνουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν ίσα δικαιώματα για όλους. I'm sorry. Συγγνώμη. Υπήρχε μια διαδικασία ε, αιτήματο ε, μετάθεσης της αναβολής της ε, ψηφοφορίας. Ο, η κανονική διαδικασία και ο κανονισμός προβλέπει μια ομιλία υπέρ, μια ομιλία με τοποθέτηση κατά. Τώρα, εντάξει, αν θέλετε να ακούσουμε και άλλες αιτιολογίες και άλλη επιχειρηματολογία, εντάξει, αλλά είναι ανώφελο γιατί ούτως ή άλλως ακούσαμε για το συμβιβασμό, ακούσαμε για τις τροπολογίες, ακούσαμε για, για μια μια μακρά, για ένα μακρύ κατάλογο. Ναι, έχετε κάτι άλλο. Όχι. Θέλω να πω το εξής. από ό,τι φαίνεται υπάρχει και ένα από ό,τι φαίνεται νέο, υπάρχει και ένας νέος συμβιβασμός ο οποίος δεν αποτελεί καθόλου συμβιβασμό ε, είναι μια πρόταση της εισηγητρίας ε, της τελευταίας ε, στιγμής που δίνει την δυνατότητα να ψηφιστεί από την τελευταία στιγμή ενώ δεν είχαν τη δυνατότητα οι πολιτικές ομάδες να μελετήσουν την τροπολογία αυτή. Μόνο εσείς αποφασίσατε ότι μπορεί να προχωρήσει η τροπολογία αυτή. Πρόεδρος, θα ακούσαμε όλες τις, όλα τα επιχειρήματα, επομένως τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε ποιος είναι υπέρ της μετάθεσης εσείς της ε, ψηφοφορίας. Κατά. Απορρίπτεται, ε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ε, ένας παραπανήσιος από το ΕΛΚ. Ωραία, πέρασε τις ψηφοφορίας. Απερίφθη το αίτημα. So we proceed to voting. Προχωράμε λοιπόν. I've told that I don't know why we have to vote μου λένε ότι πρέπει να ψηφίσουμε πρώτα το συμβιβασμό ή Δεν ξέρω γιατί. Α, so first A, sorry. Α, το A πρώτα. Ωραία, ωραία. Συμβιβασμό A, υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τώρα συμβιβασμό E, υπέρ. E, E, E.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 Περνάμε τώρα στο συμβιβασμό B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, συμβιβασμό C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός F Το ψηφίσαμε το D. Συμβιβασμός F υπέρ. Α, ναι, έχει διάφορα τμήματα λοιπόν. Ε, πρώτο τμήμα του F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβασμός H σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός I υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 183 υπέρ, κατά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 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 212 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 213 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 216 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβασμός K υπέρ κατά αποχές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 αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός εν ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 295 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 299 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 300 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, ΙΜΚΟ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ΙΜΚΟ 3 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, ΙΜΚΟ 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός ΟΟΥ σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός π σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 319 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 364 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 367 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 368 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παρακαλώ πολύ να σηκώνετε τα χέρια σας. Συμβιβασμός S σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός T σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 494 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στη συμβιβασμός β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλ 10 υπέρ κατά αποχές Έμπλου 13 σε τρία τμήματα. Υπέρ, το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έμπλου 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική X σε δύο τμήματα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 446 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται.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 Παρακαλώ να ψηφίσετε. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 502 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική AD υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 521 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 522 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5.23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5.24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ΑΕ e, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AF σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο βήμα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 446 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 551 υπέρ Α, εκπίπτει. Συμβαστική AG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AH υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική AI υπέρ. Α, έχασα τις πίσω μου σελίδες. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται συμβαστική AJ υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται Συμβαστική AK υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 11 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική AL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 κατά αποχές εγκρίνεται AQ συμβαστική πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική AR πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική AS υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική AT σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AU υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AV υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική BFA υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 709 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική AW υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AX υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AY υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική AZ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 758 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική BA υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική BB υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική BC υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική BD υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική BE υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική BF υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική BG υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική BH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική BI πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 819 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 820 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο, έτσι δεν είναι. Τσεκ, έλεγχος είναι 820, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται συμβαστική BP υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική BQ πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. συμβαστή BR υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. BL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. imco G υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική BS. Εδώ υπάρχει προφορική τροποποίηση από τους πράσινους. Ψηφίζουμε πρώτα την προφορική τροποποίηση υπέρ κατά απόχες. Μπορούμε να την ψηφίσουμε και θα απορριφθεί. Αλλά κάναμε περίπου 70 ώρες διαπραγματεύσεων για να περιλάβουμε αυτές τις λέξεις Κάπου πελήθηκαν, κάπου δεν πελήθηκαν. Τώρα ξαναγυρίσουν. Θα ήταν πιο σαφές να πω όχι στην προφορική τροπολογία που ήταν στοιχείο 70 ωρών διαπραγματεύσεις. Οπότε εσείς αντιτίθεστε. Ναι, θα ήταν σωστό. Γιατί το έχουμε συζητήσει. Χρειάζομαι τέσσερις βουλευτές να αντιταχθούν στην ψήφιση αυτή. Εντάξει, ωραία. Ψηφίζουμε τη συμβαστική χωρίς την προφορική τροποποίηση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική BK υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική BM υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική BJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α, την BO. Συμβαστική BO υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα την BJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 131 με προφορική ναι. τραπολογία υπέρ Ένσταση, ένσταση στην προφορική τροπολογία. Τέσσερα άτομα. Σηκώνουν τα χέρια του. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ναι, πολύ ωραία. Ωραία. Ψηφίζουμε λοιπόν το κείμενο χωρίς την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Έλεγχο ζήτητε. Για την 131. Ένταξη ψηφοφορία. So the vote one EPP too many. Μία ψήφος παραπάνω από το ΕΛΚ παρακαλώ. Πέρα. Απορρίπτεται. Ample A. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 132. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 133. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 134. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 135. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 136 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, ΙΜΚΟ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, Αρχικό κείμενο, λογική σκέψη 1, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 3, η, η σκέψη, η, τροπολογία 2, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, αρχικού κειμένου, ετελογική σκέψη 4, υπέρ κατά ε, εγκρίνεται Να ψηφίσουμε όλε μα τι τροπολογίε αυτέ. Δεν υπάρχει κανεί που αντιτίθεται υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, απόχέ απορρίπτεται. Αρχικού κειμένου 4 υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Η τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχέ ε, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο, η όντια υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η ιδεολογική αναφορά 13 και 14 μαζί, αν συμφωνείτε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο 15 ε, υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Η 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο τροπολογία, η τροπολογική αναφορά μάλλον 16 ε, λέει ο Πρόεδρος υπέρ. Αρχικό κείμενο, η τροπολογική αναφορά 16 υπέρ κατά Έλεγχος παρακαλώ, αρχικό κείμενο, ε, λογική αναφορά 16. Πέρασε τη εγκρίνεται. Αυτό ήταν το αρχικό κείμενο λογική να 16, 12 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο 17 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Η τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται αρχικό κείμενο, τελική αναφορά 19 υπέρ, κατά. Αρχικό κείμενο, τελογική αναφορά 19. Είστε όλοι υπέρ, υποθέτω. Αρχικό κείμενο της τελογικής αναφοράς 19. In favor, I think I see. Okay, in favor, against abstentions adopted.